Καθίστε συνάδελφοι παρακαλώ. La séance est ouverte. Άρχεται η συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι στη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7 Φεβρουαρίου στην μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολιετές δημοσιονομικούς πλαισίου δεν συζητήθηκε. Η επιφύλαξη της Ιταλίας δεν ήρθε, επομένως τα σημεία 13, 14 και 15 που ε, έχουν συνεισηγητές ε, το η κυρία Τομέ και τον κύριο Χόλπιτς, ε, αναβάλλονται τα σημεία 18 και 19 της κυρίας Γκαρδία Θαμπάλ θα συζητηθούν στο τέλος του πρωινού. Σας ζητώ επίσης να σημειώσετε ότι επειδή η Μόνικα Χόλμαγερ, η συγγήτρια, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Το σημείο 6 θα συζητηθεί μετά το σημείο 8 και 9 και θα στραφεί η σειρά του 8 και του 9. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, ε, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη ως τροποποιήθηκε. Να σας πω επίσης ότι στις 12 παρατέταρτο θα πρέπει να φύγω, αν δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας, διότι η διάσκεψη των Προέδρων θα συναντήσει τον Μάριο Μόντι ε, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους και πρέπει να παρευρεθώ εκεί ως πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών. Και τώρα να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των συντονιστών για, που ελήφθησαν συνεδρίαση της 8 Φεβρουαρίου. Αποφασίστηκε να υπάρξει μια γνωμοδότηση στην έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Απασχόλησης για την έκθεση εφαρμογής της ε, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων βάσει του άρθρου 53 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κάποια στιγμή συζητήθηκε το άρθρο 54, αλλά ε, η, ο εισηγητής θεωρεί ότι το άρθρο 53 είναι το κατάλληλο. Αποφασίστηκε επίσης να ζητήσουμε την έγκρισή σας για να υπάρξουν δύο εκθέσει πρωτοβουλία για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και τους ίδιους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεισηγητέ ε, η Ζαμπέλ Τομά και ο Γιάννη Όλπριχτ και ε, για τους ίδιους πόρους Γιάννου Λεβαντόφσκι και Ζεράρ Ντεπρέ. Τέλος, αποφασίστηκε να εγκρίνουμε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της έκθεσης ε, για την ε, κατάσταση δαπανών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2018 που πρότεινε ο κύριος Άσουαρτς, ο εισηγητές. Η παρουσίαση θα γίνει στις 6 Μαρτίου, 15 Μαρτίου 12 η ώρα οι τροπολογίες, δεύτερη ανταλλαγή από 20 Μαρτίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Πλοϋπολογισμών στην Ολομέλεια του Απριλίου. Βεβαίω μπορεί να υπάρξουν προθερμογέ στο χρονοδιάγραμμα λόγω του χρονοδιαγράμματο του Προεδρείου, το οποίο θα επιβεβαιωθεί αργότερα. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίε. Σα παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες σας στι συσκευέ. πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση του συναδέλφου Νέτσμι για το τομέα προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. για την υπόθεση Trend Over the Retail στις κάτω χώρες. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να δούμε έναν έλεγχο πρώτα. 23 κάρτες, 22 ψήφοι. Κύριε Ταράου, η κάρτα σας δεν δούλεψε. Ε, ε, Εντάξει, δουλεύει. Ωραία. Παράγραφος 7, τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Είναι εκτός πεδίου. Επομένως, ε, μη παραδεκτή. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και για το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Και τώρα έχουμε μια μεταφορά που χρειάζεται και την ε, ε, γνωμοδότηση του Γενικού Εισηγητή του κ. Γκάιερ. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχε πάρα πολύ κίνηση σήμερα το πρωί στη γειτονιά μου και γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη, καθυστέρησα. Η μεταφορά την οποία και σας προτείνω, είναι η ψηφοφορία που κάναμε. Θα έχει μια λογική συνέπεια. Ε, Οφανθήκαμε θετικά για τις προτάσεις προκειμένου από το, παγκοσμιο... από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι. Αυτός είναι ο λόγος της μεταφοράς, την οποία και σας ζητώ να εγκρίνετε. Pardon, le vote est un vote électronique. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Le scrutin est clos. ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Monsieur sur les autres sections, Ο κύριος Ταράν για τις άλλες ε, κατηγορίες δεν υπάρχει έτοιμα μεταφοράς. Σας έχουν ζητήσει τίματα μεταφοράς. Δεν υπάρχουν κύριε Ταρά. Ωραία. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία, αλλά θα συνεχιστεί μόλις έρθει η Μόνικα Χολμάιερ για ε, τα κτίρια. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στο Σίκφριτ Μουρεσάν, το Γενικό Εισηγητή μας, ο οποίος ε, θα μας ε, παρουσιάσει μια πρώτη εικόνα για τον προπολογισμό του 2018. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα το πρωί θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την κατεύθυνση προς την οποία θα οδηγήσουμε τον προϋπολογισμό της Ένωσης το 2018. Εγώ σας έχω ήδη στείλει μία πρόταση ψηφίσματος για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό μας το 18. Δηλαδή στην ουσία ένα κατάλογο προτεραιοτήτων πολιτικών. Ε, υπάρχει δυνατότητα τροπολόγησης και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 6 Μαρτίου και στην κανονική Ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο. Είναι μια ευκαιρία να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν καταθέσουν την πρόταση προϋπολογισμού το μήνα Μάιο, να μας εξηγήσουν το πώς προτείνουν να χρησιμοποιήσουν τους σχετικά περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να κάνουν αυτό το οποίο επιθυμούν οι πολίτες της Ευρώπης. Πιστεύω και αυτή είναι η βασική μου γραμμή, αν θέλετε, για το 2018, Νομίζω ότι αυτό το οποίο περιμένει ο Ευρωπαίος πολίτης είναι ανάπτυξη, θέσεις απασχόλησης σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια περάσαμε εποχές περίεργες και πάρα πολύ ενέργεια θα έλεγα δόθηκε στις συζητήσεις μας για τα δημοσιονομικά ε, για το θέμα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, θα πρέπει όμως να στείλουμε και το μήνυμα ότι εμείς δεν ξεχνάμε τις παραδοσιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η κάλυψη των αναγκών των λαών της Ευρώπης στον τομέα της απασχόλησης. Θέσεις απασχόλησης κοινωνικά βιώσιμες, ικανοποιητικές και σωστά αμοιβόμενες. Η οικονομία θα το καταφέρει αυτό και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, να επενδύσουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες, να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες και με το Horizon 2020 και με το COSME και με το Connecting Europe Γνωρίζουμε καλά ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, λειτουργεί με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε το ποσοστό των προγραμμάτων τα οποία ζητούν χρηματοδότηση έχει φτάσει μόνο στο 12%. Στις 100 αιτήσει 12 δεκτές. Το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί τα προγράμματα καινοτομίας όπως επίσης και το Connecting Europe δεν μπορούν να στηρίξουν όπως επιθυμούσαμε ε, τις προτάσεις ε, οι οποίες είχαν κατατεθεί λόγω της δημιουργίας κυρίως του στρατηγικού επενδυτικού ταμείου. Συνεπώς λοιπόν το μήνυμα για το 18 είναι ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες ότι θα στηρίξουμε την πραγματική οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης σταθερών και κοινωνικά αποδεκτών. Φυσικά η προσφυγική κρίση είναι εδώ, αλλά η οικονομική κατάσταση είναι κάτι το οποίο απαιτεί φροντίδα, δεν πρόκειται να βελτιωθεί αυτής. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε λοιπόν ακόμα περισσότερο το γιούρο Υπάρχουν εδώ βέβαια και αρκετά θέματα τα οποία δεν άπτονται του προϋπολογισμού της Ένωσης, αλλά και μέσω του προϋπολογισμού θα πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομία. Τώρα για συγκεκριμένα θέματα όπως το ΕΦΣΥ που ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια. Είναι μια καλή προσπάθεια και θα θέλαμε να συνεχιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στον τομέα της προσθετικότητας όπως και στον τομέα της γεωγραφικής διανομής, διασποράς. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν και με άλλες πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων η οποία παραμένει βελτιώσιμη έτσι ώστε στο τέλος να δημιουργηθούν ικανοποιητικές θέσεις απασχόλησης σωστά αμοιβόμενε για τους ευρωπαϊκούς λαούς και να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πρόγραμμα Εράσμους. Η πολιτική συνοχής είναι μια βασική πολιτική που θα χαρακτήριζα πολιτική επενδυτική και η περιγραφή η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση Μόντι είναι καλή γιατί χρησιμοποιεί την πολιτική συνοχή σαν μια πολιτική μέσα από την οποία ωφελούνται όλοι, όχι μόνο οι χώρες καθαρής συνεισφορής. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του juste retour της δίκαιης επιστροφής, όπως ακριβώς το προτείνει ο κύριος Μόντι στην έκθεσή του στην οποία πήραμε και εμείς μέρος. Οικονομία λοιπόν, απασχόληση από τη μία, ασφάλεια όμως από την άλλη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο, ο κόσμος, οι πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς και οι επιχειρήσεις δεν νιώθουν ασφαλείς και δεν διευρύνουν την οικονομική τους δραστηριότητα όταν υπάρχουν προβλήματα ανασφάλειας. Ξέρουμε ότι οι πόροι στο τρίτο τμήμα είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα άλλα μέσα γιατί το, MF, το, διεθνές, το πολιετές συγγνώμη, δημοσιονομικό ε, δεν ήταν ικανό το 2013 όταν δημιουργήθηκε να προβλέψει την εξέλιξη των πραγμάτων. Τίθεται λοιπόν το θέμα της χρήσης των περιορισμένων πόρων τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης, στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και για να μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε την αίσθηση ασφάλειας του πολίτη και να δαπανίσουμε τα χρήματα φυσικά που έχουμε διαθέσιμα, αλλά δυστυχώς ε, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερα πάντα στον τομέα της ασφάλειας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στην γειτονία μας, στην Ανατολική και στην Νότια. Πέρυσι είχαμε πάει με συναδέλφους στον Λίβανο, στην Ιορδανία, επισκεφθήκαμε πρόσφυγες. Είναι χώρες αυτές που δέχθηκαν ένα εκατομμύριο μετανάστες η καθεμία. Και είδαμε ότι πολλά μπορεί να γίνουν με την στήριξη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Είναι ευθυνότερο να στηρίζει κανείς τους πρόσφυγες κοντά στη χώρα προέλευσής τους και όχι στην Ένωση. Και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες εφαρμόζουν επιτόπου τα προγράμματα, αναγνωρίζουν ότι δεν θα ήσαν σε θέση να στηρίξουν, να παρέχουν τρόφιμα, πόσιμο νερό στους πρόσφυγες της περιοχής, αν δεν είχε προϋπάρξει η δική μας υποστήριξη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες, τις ουσιαστικές της μετανάστευσης και των προσφυγικών ρευμάτων. Τα χρήματα τα οποία δαπανάμε επί τόπου νομίζω ότι είναι χρήματα τα οποία είναι ε, σωστά επενδεδημένα. είναι χρήματα τα οποία ελέγχουμε σωστά, ε, αποτρέπουμε την κατάχρηση των πιστώσεων αυτών, αποτρέπουμε τις απάτες, καλύπτουμε τις ανάγκες των δικαιούχων και πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υγεία, στην εκπαίδευση σε αυτές τις χώρες που είναι σχεδόν γειτονικέ για μας έτσι ώστε οι συνθήκες ζωής, οι συνθήκες διαβίωσης να βελτιωθούν και η ανάγκη μετανάστευσης να μειωθεί. Λοιπόν, οι πληρωμέ είναι σημαντικές για τον επόμενο χρόνο. Το ποσοστό απορρόφησης στα δύο πρώτα χρόνια της περίοδου 13-16 ήταν χαμηλές. Ελπίζουμε τα λειτουργικά προγράμματα να αποκτήσουν υψηλότερη ταχύτητα από το 18 και το 19. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκή σπόροι, γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Όταν προτάθηκε η συγκεκριμένη έκθεση δεν είχαμε την πρόταση του Συμβουλίου για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού. Αυτή την εβδομάδα έγινε μια πρώτη συζήτηση αλλά δεν έχει υπάρξει καταληκτική τουλάχιστον πρόοδος. Εάν λοιπόν το πρώτο που θέλω να πω μάλλον εδώ είναι ότι αποφασιστεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού και θα επηρεάσει το 18, τον προϋπολογισμό του 18, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία τις επόμενες εβδομάδες αλλάξουν και εφόσον χρειαστεί τα στοιχεία αυτά να ανταλάβουμε υπόψη μας για τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτό μπορεί να γίνει μέσω των τροπολογιών. Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού και εφόσον υπάρξουν κάποιες προτάσεις από εκεί θα ε, παίξουμε και εμείς τον υποστηρικτικό μας ρόλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε με προσοχή. Ε, προσβλέπω στην δική σας συμμετοχή και ε, περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων κατά τη διάρκεια των επομένων ημερών. Ευχαριστώ τον γενικό εισηγητή μας, που μας έδωσε τις προτεραιότητες του για το 2018. Θα προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης πρώτα, μετά στους συντονιστές που έχουν ζητήσει το λόγο και τέλος τα μεμονωμένα μέλη που έχουν ήδη εγγραφεί. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη εγγραφεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή, τον κύριο Μούρεσαν, για το κείμενο το οποίο μας υπέβαλε, αλλά και για την ε, πολύ καλή συνεργασία για το, είναι, για το 2018 και τον προϋπολογισμό. Βρισκόμαστε σε πολύ, καλή δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο από αυτή την πλευρά και ελπίζω και για το περιεχόμενο. Να περάσω τώρα στην ουσία αυτών των οποίων μας υπέβαλε, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ισορροπημένο όσον αφορά τη στήριξη στην ε, απασχόληση των νέων και ε, στο σημείο που ζητά αύξηση για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, την βασική έρευνα τη θεμελιώδη έρευνα. Πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και να ζητάμε κάποια πράγματα, να μην έχουμε απλώς ε, διατήρηση των ποσών που έχουμε στο κόσμο. Ε, θα τα αναφέρω επιγραμματικά ανατίτλους. Επίσης, ε, πολύ καλή η πρόταση για την εγγύηση για την νεολαία, αλλά έχουμε και κάποιες αμφιβολίες, τις οποίες έχουμε εκφράσει επανειλημμένως, για το Interrail, και το αναφέραμε και ως πολιτική ομάδα άλλωστε αυτό, εμείς ε, τίνουμε μάλλον προς ένα ολοκληρωμένο πρόβλημα για την ε, πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό και ε, να μην τους δίνουμε απλώς ένα εισιτήριο τρένου για τις διακοπές τους. Βέβαια θα τα συζητήσουμε αυτά. Όσον αφορά τις εσωτερικές προκλήσεις, συμφωνούμε στη δέσμευση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ασφαλείας, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την προσπάθεια για την υποδοχή ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου και να έχουμε μια προστασία των συνόρων που δεν θα πρέπει να θεωρείται όμως από τη στενή έννοια της ασφάλειας και μόνον. Η αίσθηση της ασφάλειας είναι να έχουμε ένα όραμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα είναι κοινωνικό, πολιτικό και γεωπολιτικό για το μεταναστευτικό φαινόμενο. Όσον αφορά τις εξωτερικές προκλήσεις, συμφωνώ μεν ως προς την ανάγκη να σταθεροποιήσουμε τις πιο πιεστικές κρίσεις στην Ουκρανία και στη Λιβύη, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και τα διαρθρωτικά μέσα στην ανάπτυξη και στη συνεργασία. Πολύ καλά υπενθυμίζεται στο κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε στο νέο καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια μέσα που έχουμε ήδη στο τίτλο 4 του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις τεχνικές ε, δομές του προϋπολογισμού, Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναφορά στη δημιουργία ένα πραγματικό σύστημα ίδιων πόρων, που είναι κάτι το οποίο ούτω ή άλλω προωθούμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα και σε ένα κείμενο σαν αυτό το οποίο συζητούμε τώρα. Όπως επίσης και ως προς την ανάγκη να ε, δούμε αμέσω τι θα γίνει με το θέμα του Brexit και τους λογαριασμούς εκεί. Να μην βρεθούμε ξαφνικά στον προπολογισμό με προεκπλήξεων και ε, να έχουμε αντιμετωπίσει ε, εντάσεις και δυσκολίες εκεί. Και επίσης να αναφερθώ επιγραμματικά και στα όσα λέτε για την πολιτική συνοχή. Συμφωνούμε και με αυτά. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι Ο, η κατεύθυνση που ακολουθείτε είναι θετική, αλλά ως σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, έχουμε κάποιες απόψεις, θα τα προωθήσουμε, ίσως θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες για τα ε, θέματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Κυρίως θα επικεντρωθούμε σε αυτά και ε, στους τίτλους 3 και 4. Νομίζω ότι θα δούμε και κάποια πράγματα ως προς τη διατύπωση ε, ίσονα σημασίας. Όπως έλεγα, θεωρώ ότι ξεκινάμε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια προσπάθεια να επιδείξουμε λίγο μεγαλύτερο στένους και να έχουμε ένα ακόμα πιο φιλόδοξο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλμελ για το ECR. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς να ευχαριστήσω τον Ζίγκφριντ είναι πραγματικά πολύ ισορροπημένη η έκθεση. Πολύ καλή. Θα ήθελα να ενισχύσω κάποια σημεία και ενδεχομένω να προσθέσω και κάποια άλλα. Καταρχά, δικαίω επεσήμανε ότι θα πρέπει να απασχολήσουμε και να εμπλέξουμε πιο πολύ τον πολίτη. Ο πολίτη θα πρέπει να καταλάβει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνουμε με τα χρήματά του. Δεν είναι δικά μα τα χρήματα αυτά. Εμεί είμαστε απλά διαχειριστέ των πόρων αυτών. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε πραγματική επικουρικότητα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε, θα πρέπει να ενεργούμε μόνο αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από ό,τι τα κρατημέλη. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα που μας απασχολούν και εμένα προσωπικά, για παράδειγμα στην κλιματική πολιτική η κοινή δράση, γιατί η πολιτική για το περιβάλλον, για το κλίμα ε, είναι τομείς όπου μπορούμε πολύ καλύτερα να δράσουμε ως σύνολο παρά ως ε, μονάδες. Και στην ενεργειακή πολιτική πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά σημεία όπου τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν στις δράσεις τους και σε τελική ανάλυση να πετύχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα από το καθένα κράτος μόνο του οι κλιματικές ισορροπίες, οι γεωγραφικές ισορροπίες ε, στα κράτη-μέλη είναι εντελώς διαφορετικές και δεν μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε μία μέθοδος, ε, μία μέθοδο που να ισχύει κατά αποκοπήν για όλους. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ενώσουμε τις δυνάμεις ε, όλων των κρατών μελών για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που θα είναι επίσης καθοριστικό είναι να επιδείξουμε τόλμη, αλλά όχι τόλμη μόνο για να κάνουμε τυφλά όλο και πιο πολλά μαζί, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε αντιθέτω στο τι μπορεί να κάνει πραγματικά καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια πράγματα είναι αρμόδια και πού θα πρέπει να μην εμπλακεί καθόλου. Γιατί σε τελική ανάλυση δεν πιστεύω ότι ήταν καλή η λύση το να ψάχνουμε και να ξεψαχνίζουμε προβλήματα για να προσπαθεί η Ευρώπη να καταρτήσει πρόγραμμα για τα πάντα. Γιατί έτσι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση και αδιαφανή και άδικη στην τελική ανάλυση. Γιατί κάπου κάποια προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν και κάποια άλλα όχι. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια λιτή Ευρώπη. Και θα πρέπει να φροντίσουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα πετυχαίνουμε να είναι μετρήσιμα και αποτελεσματικά. Εγώ είμαι μεγάλος υπερμαχό τη ε, πολιτική συνοχή, αλλά να είναι και επιτυχής η πολιτική συνοχή Αλλιώς τι πολιτική συνοχή είναι. Δηλαδή. Αν δίνούσε κάποιον για 10-20 χρόνια χρήματα και στη συνέχεια έχουμε την εντύπωση ότι δεν πετύχαμε κάτι συγκεκριμένο, απλά πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε κάποιο έργο, τι έχουμε πετύχει. Ίσως έχει έρθει η ώρα να τα αμφισβητήσουμε αυτά και ίσως αν κάποιος άλλος έχει μια καλύτερη ιδέα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η καλύτερη ιδέα. Κάτι τελευταίο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερως είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Η κρίση μεταναστευτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θυμάστε. Κάποιο είπε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε και τρόπους για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της μεταναστευτικής κρίσης. Εγώ είπα και το έλεγα πάντα ότι τα χρήματα δεν αρκούν για το σκοπό αυτό. Χρειαζόμαστε μια σωστή στρατηγική και μάλιστα ολοκληρωμένη από το Α μέχρι το Ω ή ιδάλω. Οτιδήποτε και να κάνουμε είναι αυθαίρετο. Αυτή η στρατηγική λοιπόν, λοιπόν δεν, δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν ε, διάφορε προσεγγίσει. Δεν είναι απαραίτητα εσφαλμένε, αλλά χρειαζόμαστε ένα συνολικό σύστημα. Συνθήκη του Δουβλίνου και όλα όσα συγκαταλέγονται σε αυτά. Τα ξέρετε άλλωστε όλα αυτά αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα αποσπασματική η δράση μας και δεν ε, μας, μας προχωράνε και μας ε, κινούν, μας υποκινούν οι εξελίξεις πιο πολύ. Πρώτα θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική και μετά νομίζω ότι δικαιούμαστε να καταρτήσουμε και να ε, δαπανίσουμε κονδύλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γιατομάκη. Ζήτησε συγγνώμη, δεν θα πάρει το λόγο η κυρία Νίριατα, εάν είναι παρούσα στην έτωση. Ο κύριος Ταράμ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να επενέσω τον εισηγητή για τις προκαταρτικές αυτές οι ιδέες που μας επέβαλε. Είναι καλό το έγγραφο για να αποτελέσει βάση της μελλοντική συζήτησης. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε μια μικρή, μικροσκοπική ομάδα, αλλά σημαντική ομάδα των πρασίνων στο Κοινοβούλιο. Και πάντα μας απασχολεί αυτή η πράσινη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Ίσως λοιπόν το σημείο, η έλλειψη στην οποία αναφέρομαι στην παρούσα είναι η δυνατότητα να προωθηθεί σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή η πράσινη μετάβαση, η συνοπτική και συνεκτική πράσινη μετάβαση. Αυτό δεν τονίζεται παρκώς, πιστεύω, στο κείμενό μας. Θα κάνουμε λοιπόν κάποιες τροπολογίες και για το θέμα το οποίο αναφέρατε και το οποίο σχετίζεται και με τη μεταναστευτική κρίση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε από κοινού να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ των όσων χρειαζόμαστε για την ασφάλεια και των ε, θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχουν καθοριστεί από την δεκαετία του 50 σε διεθνές επίπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε και κάνετε αναφορά στη μεταρρύθμιση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά για μένα το καλύτερο κομμάτι του κειμένου και το χειροκροτώ είναι το σημείο 55 που τονίζει τη σημασία του Κοινοβουλίου σε θέματα προπολογισμού ως το μοναδικό αιρετό όργανο από τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ που το προσθέσατε. Ευχαριστώ κύριε Ταρόν, λέει ο πρόεδρος. Η EFTD. Ποιος είναι ο συντονιστής από το EFTD? Ο Σκιώτη, συγγνώμη. Ο κ. Ζόλτεκ από το ΙΕΝΕΦ. Επιτρέψτε μου να αντικαταστήσω την κυρία Γιάτεν για να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις ε, για την πολιτική μου ομάδα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μουρεσάν για την πρώτη του έκθεση. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό το οποίο χρειαζόμεθα όλοι είναι μια στρατηγική αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και εσείς έχω πάει πολλές φορές σε επιτόπου σε περιοχές όπως η Ορδανία και ο Λίβανος. Έχω πάει στην Γάζα, στην Υπεριορδανία, Παλαιστίνη και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση όταν είμαι επιτόπου είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτό που θα ονόμαζα ένας οδικός χάρτης. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν ήσαν σαφείς. θα βέβαια παρόντες, θα η πρώτη δωρήτρια δύναμη στην Παλαιστίνη, αλλά αυτό δεν φαίνεται κάπου. Και όταν γίνεται μια ειρηνευτική πολιτική συνάντηση, είναι παντελώς απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι παράδοξο. Είμαι θα η πρώτη δωρήτρια δύναμη όπως είπα, αλλά η πολιτική μας διάσταση ελείπει. Συνεπώς, ως εκπρόσωποι της επί του προϋπολογισμού αρχής. Νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στους κυβερνήτες, όποιοι και αν είναι αυτοί, να διευκρινίσουν το όραμα και τις προτεραιότητες, διότι τι άλλο είναι ο προϋπολογισμός από τη μεταφορά ε, στην πρακτική ε, εφαρμογή των ιδεών. Αν δεν υπάρχουν όμως ξεκάθαρες ιδέες, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, απλά παρατείνουμε τις διάρκειες παρεμβάσεων προσπαθούμε να καλύψουμε δαπάνες με χρήματα τα οποία είναι δυστυχώς λιγότερα από όσα χρειαζόμεθα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ανεργία των νέων, η κινητικότητα των νέων, το έρασμος. Το έρασμος ε, ε, μιλά στους Ευρωπαίους, τους νέους Ευρωπαίους. Όταν ρωτάνε τους Ευρωπαίους τι συμβολίζει την Ευρώπη, πρώτα λένε βέβαια το ευρώ και μετά το έρασμος. Συνεπώς λοιπόν, εγώ δίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την μαθητεία, την κατάρτιση και για τους εργάτες και για τους μηχανικούς και ε, βλέπω ότι στις χώρες που υπάρχει ε, παράδοση στον τομέα της μαθητείας όπως η Αυστρία και η Γερμανία ε, δεν υπάρχει ανεργία στους νέους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Φυσικά η μετανάστευση και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και παραμένει σημαντικό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη. Είναι μείζον το θέμα διότι από ό,τι φαίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες πιθανώς να υπάρχει μια στροφή σιγά σιγά στον τομέα αυτό ε, και να βαδίζουν προς μια κάποια μορφή απομονωτισμού. Αυτό θα ήταν ένα σοκ για την Ευρώπη. Τώρα για τον κύριο Τάραντ, ε, όπως είπε και ο κύριος Τάραντ, ε, για την ενεργειακή μετάβαση. Σαν παράδειγμα η κατασκευή ηλιακών πινάκων ε, προφανώς θα πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Από την άλλη όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε το dumping το οποίο ε, ασκείται μέσω της εισαγωγής κινέζικων προϊόντων. Και διάφοροι λέγουν τώρα ότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήσαν κατά της λήψης αμυντικών μέτρων που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι πράγματι παράδοξο. Εφόσον θέλουμε να διασώσουμε την απασχόληση, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι κάναμε για το χάλιβα. Αυτό το οποίο κάναμε φαίνεται ότι λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο. Ίσως θα πρέπει να επεκταθεί και εις άλλες δραστηριότητε και να διατηρήσουμε, να διασώσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Απαιτείται και το κατάλληλο διακανονιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά τώρα κάποιοι συντονιστές που δεν μίλησαν μέχρι τώρα θα ήθελαν το λόγο ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Να τον συγχαρώ γιατί είναι σαφείς οι προτεραιότητες ε, που μας παρουσίασε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ανάπτυξη, σύμφωνη, χρειάζεται πιο πολλέ θέσει απασχόληση. Οι πολίτε πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια. Και η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί αργά ή γρήγορα από πλευρά χρηματοδότηση και προπολογισμού. Επίσης επισημαίνει ότι προσοχή χρειάζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις νέους. Θα πρέπει ενισχύσουμε το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Erasmus Plus αποτέλεσε πάντα μία από τις προτεραιότητές μας. Το θέμα του Ιντερελ έχει ήδη περάσει στην Ολομέλεια με την υποστήριξη του μεγαλύτερου τμήματος των πολιτικών ομάδων. Είναι συμβολικό μεν στη σημασία του, αλλά πάρα πολύ ουσιώδες σε ό,τι αφορά αυτή την αίσθηση του ανήκειν ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προωθεί ακριβώς την επαφή με τις άλλες χώρες. Και τις αξίες μας. Θα ήθελα να, υποσ... να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι μιλάμε για μια χρηματοδότηση που αντιπροσωπεύει το 1% του εθνικού ΑΕΠ. Με αυτό το 1% προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Και η επίδραση του προϋπολογισμού αυτού δεν είναι πάντα σαφής. Δεν αντιλαμβάνονται πάντα οι πολίτες τι ακριβώς χρηματοδοτείται, τι ακριβώς επιτυγχάνεται. τα σχολεία που χτίζονται, οι κατοικίε. Και όλα αυτά για τα οποία ευθύνεται ο προϋπολογισμός. Είναι σημαντικό λοιπόν τα προγράμματα όπως το πρόγραμμα το 2020 για την έρευνα για να γίνει πιο σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το 1% λοιπόν του Εθνικού ΑΕΠ πετυχαίνουμε πολλά. αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά συνείδηση και ενημέρωση γι' αυτό. Και το γεγονός ότι το 6% μόνο του προϋπολογισμού αυτού ε, προορίζεται για διοικητικά έξοδα. 94% λοιπόν του προπολογισμού είναι χρησιμοποιείται για επιδετικούς σκοπούς. Η προβολή λοιπόν του γεγονότος αυτού είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φροντίσουμε. Επίσης, να φροντίσουμε οι προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι είναι κάτι το οποίο τα κρατη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κρατη από μόνα τους τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από το προσφυγικό, από το μεταναστευτικό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό πάρα αυτά, γιατί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι άλλη μια αναπαλωτρίωτη αξία και ξέρουμε ότι θα πρέπει να πολεμήσει για αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από κοινού. Η καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφύγης επίσης προαπαιτεί αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς ε, η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση και η πρόληψη αυτής επίσης μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες τις υποστηρίζω. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο προπολογισμό είναι περιορισμένος, με τον οποίο ως τώρα έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με τις οποίες έχουμε έρθει αντιμετωπί και να δώσουμε απαντήσεις στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το ότι συχνά η ανταπόκριση αυτή, η απάντηση αυτή που δώσαμε δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε. Και ασφαλώς θα πρέπει να διαχειριστούμε και τις προσδοκίες του καθενός. Δεδομένου του προπολογισμού των κρατών μελών που αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, τον είπα για παράδειγμα, Αυτό δεν σημαίνει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ απλά δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα με τον διαθέσιμο προπολογισμό και σίγουρα οι πληρωμέ θα αποτελέσουν ένα πρόβλημα. Ελπίζω, και αυτό υπόθηκε ήδη, ότι δεν θα πρέπει να βγάζει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα από το γεγονός ότι από την πολιτική ε, συνοχή έχουμε ακόμα 13 δισεκατομμύρια τα οποία που δεν έχουν απορροφηθεί. Μεγάλο τμήμα πηγαίνει για την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία. Άρα θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τα θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη για να επιταχυνθεί επιτέλους η πολιτική συνοχή και να μην υπάρχουν προβλήματα. τα οποία έχουν επιστημωθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το θέμα των πληρωμών είναι θέμα αξιοπιστίας, επαναλαμβάνω θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και να πληρώσουμε τα χρωστούμενα. Οι δεσμεύσεις αυτές δε, και οι αλλαγές στις πληρωμές είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Για τις καθυστερήσεις, για παράδειγμα, στις πληρωμές. Προφανώς αυτό η καθυστέρηση οδηγεί σε τοκισμό Άρα, θεωρώ ότι στον προπολογισμό οι προτεραιότητε είναι εξαιρετικά σαφεί και οι πολιτικέ ομάδε θεωρώ ότι συμφωνούν με αυτέ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρδιά Θαμπάλ. Δεν θέλω το λόγο. Ούτω ή άλλω ο συνάδελφο εξήγησε πάρα πολύ καλά την θέση τη ομάδας. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος από τους συντονιστές που θέλει το λόγο. Νομίζω ότι είπαν ε, αυτά τα οποία επιθυμούσαν. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα με προσοχή και εγώ το έγγραφο του συναδέλφου του Ζίκφριντ και νομίζω ότι προκειμένου να πετύχουμε την ισορροπία την οποία επικαλέστηκαν πολλοί, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάποια σημεία, τα οποία θα έπρεπε να αναφερθούν. Να συμφωνήσουμε τι πρέπει να αναφερθεί. Χριστιανοδημοκράτης ε, ο συνάδελφος. Όταν ε, μιλάμε για την ανάπτυξη και την απασχόληση κτλ. Πολύ απλά μου λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να αναφέρονται και θα πρέπει να υλοποιηθούν. Ένα εξ αυτών είναι η αναφορά της κοινωνικής ε, ισορροπίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αυτή η διάσταση θα πρέπει προφανώς να προβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραπάνω και να ληφθεί υπόψη και στην χρηματοδότηση όπως και τα στοιχεία και οι πτυχές της βιωσιμότητας. Κοιτάξτε, είναι λεπτομέρειες αυτά, μικροπράγματα. Και σίγουρα ο σκιώδης μας θα υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες και εγώ με χαρά θα συμμετέχω στη διαδικασία. Αλλά πέρα από κάποιες λέξεις κλειδί που μου λείπουν και θα πρέπει να συμπεριληφθούν, θα ήθελα σε τρία σημεία ενδεχομένω να προσθέσουμε και μια προοπτική, αν θέλετε. Υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο υπαγορεύει ότι θα πρέπει η νέα ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει στην ε, ασφάλεια. Σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά βλέποντας το τι βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως θα έπρεπε να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει και άλλο η τάση αυτή και το θέμα της χρηματοδότησης τέτοιων μέτρων με ανησυχεί που δεν συζητιέται στην Επιτροπή εδώ. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι με τον προπολογισμό του 1% ΑΕΠ δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τον κόσμο. Μπορούμε να προωθήσουμε κάποιες θέσεις, να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα, ναι. Αλλά αν θέλουμε στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας να κάνουμε σημαντικά βήματα, θα πρέπει οι υπεύθυνοι προπολογισμού του Κοινοβουλίου να επισημάνουν προς όλους τους υπόλοιπους ότι πολύ απλά δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα, τους απαραίτητους πόρους. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί πιο σαφέστερα, σαφέστερα μάλλον, το σημείο αυτό. Το ίδιο πιστεύω και για τις εξωτερικές προκλήσεις. Φυσικά και υπάρχουν άλλες κρίσεις που ζητούν την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτές που αναφέρονται στο σημείο 18. Θα ήθελα να τονιστεί και η σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας και των μέσων πρόληψης κρίσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε το τι γίνεται και με τα trust funds, με τα καταπιστευματικά ταμεία, τα οποία μας προκάλεσαν πολύ μεγάλο πονοκέφαλο όταν τα συστήσαμε και τι, πώς πάνε, πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν. Και θα ήθελα να επισημάνουμε εκ νέου στα κρατη ότι θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αρκούν οι συμβολές τους και οι συνεισφορές τους στα καταπιστευματικά ταμεία. Κάποιο, ένα τελευταίο τώρα σημείο. Ίσως ε, το λάβει υπόψη και ο Ζίγκφριτ θα κάνω τροπολογία. Είναι το ΕΦΣΑΙ, το για την Αφρική. Ω ε, για τον προπολογισμό του 2017 Σα είχα αναφέρει ότι πιστεύω ότι με την επέκταση του προϋπολογισμού και με την επέκταση των στοιχείων του προπολογισμού θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και θα πρέπει σε κάποια φάση στην Επιτροπή μας να μην αμφιβάλλουμε για την ιδέα του μέσου αυτού αλλά να ενταχθούμε στην διεύρυνση του μέσου χωρίς την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου και μάλιστα από την κατηγορία από την, ε, το κεφάλαιο 4. Και αυτή η διαπραγματεύση λοιπόν για την χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ για την Αφρική θα πρέπει να ε, συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία αυτή και να έχουμε μια ιδέα για πέρα πρόκειται. Τέλος αυτό που αναφέρεται στο 24 για τον ρόλο των ίδιων μέσων. Εδώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι φεύγουν οι Βρετανοί είναι, σημαίνει ότι αφαιρείται το μεγαλύτερο εμπόδιο που είχαμε για την χρήση των ιδίων πόρων. Δεν μπορούμε πλέον να κρυφόμαστε πίσω από του Βρετανού και την δικαιολογία αυτή. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε λοιπόν και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία που θα έχουμε. Και τέλο, τον προπολογισμό για το 2018 θεωρώ δεν μπορούμε να τον συζητήσουμε χωρί να συζητήσουμε τον Brexit και τι συνέπειε που θα έχει για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι οι βαθίε αλλαγέ οι οποίε. Ε, θα σημειωθούν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν ε, σταματήσει και αφαιρεθεί ένας βασικός παράγοντας δεν μπορούν να μελεθούν. Ούτε σε ό,τι αφορά τα, τη συζήτηση για τα έσοδα, ούτε σε ό,τι αφορά τα, τη συζήτηση για τις δαπάνες. Μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Και κύριος Δενανό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή ε, που μας πρότεινε το κείμενο. Σε γενικές γραμμές πηγαίνω, πιστεύω πως πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να είναι ακόμα πιο φιλόδοξο. Ξέρουμε πώς τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Ε, μετά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου, ε, ξέρουμε ότι ε, στο αρχικό κείμενο είμαστε πολύ πιο κάτω από αυτά τα οποία επιθυμούσαμε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε είναι τις διαρθρωτικές πολιτικές, τις πολιτικές συνοχής και την ε, κοινή γεωργική πολιτική. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν απασχόληση. Και τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις, χρειάζονται υποδομές, πρόσβαση, οδικά δίκτυα, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και κυρίως ε, ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ε, δραστηριοποιούνται. Και επίση θα πρέπει να υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη για να μπορέσουν να δώσουν νέο προσανατολισμό στην παραγωγή του. Και επίση χρειαζόμαστε και εξειδικευμένο προσωπικό. Και εδώ βρίσκουμε και το θέμα τη νεολαία, τη βοήθεια προ του νέου για να αποκτήσουν εξειδίκευση, να βρουν μια εξειδικευμένη θέση εργασία και εξού και η εγγύηση για την νεολαία, εξού και το Εράσμου, εξού και πιλωτικά προγράμματα όπω αυτά τα οποία προτείνατε εσεί κύριε Πρόεδρε και πολλά άλλα πιλωτικά προγράμματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν βοηθήσουν τους νέους να βρουν το δρόμο τους. Και επίσης, ως προς τα θέματα της υποδοχής, προφανώς και πρέπει να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε ε, πρόσφυγες, αλλά δεν ε, θέλω η συμφωνία για την Τουρκία να είναι το α και το ω της συμφωνίας υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι το θέμα της άμυνας, το οποίο αναφέρθηκε επανειλημμένως, είναι ουσιώδες ε, σε, στο διεθνές πλαίσιο που γνωρίζουμε σήμερα Αφενός έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες ε, ε, αποδεσμεύονται, τη, Ρωσία που απειλεί και το Ηνωμένο Βασίλειο που θέλει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα γιατί ήταν μία από τις δυνάμεις της ε, στρατιωτικής άμυνας και η Γαλλία θα βρεθεί λίγο απομονωμένη εδώ. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε τη διάβια να σκεφτούμε τα θέματα της άμυνας όπως ε, ανέφερε και ο κύριος Γκάιερ προηγουμένως. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν, επιτρέψτε μου και την ε, έκφραση ε, απλώς έτσι φιρδινμίγδιν, θα πρέπει να δούμε ε, τι πρέπει να κάνουμε στον προπολογισμό. Πρέπει ο προπολογισμό να είναι πολύ υψηλότερος για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλα αυτά τα οποία έχει δικαίωμα να ασκήσει. Αν δεν έχουμε προπολογισμό, δεν έχουμε ίδιου πόρου, δεν χρειάζεται να κάνουμε όνειρα και να κάνουμε και μεγάλες συζητήσεις. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Αυτή είναι η διπόρη βεβαίω. Θα μπορούσε να είναι και η καταπολέμηση της απάτης. Μην το ξεχνάμε όλα αυτά. Ε, πρέπει να κάνουμε λοιπόν πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και αν υπάρχουμε έναν προπολογισμό ο οποίος θα είναι άξιος λόγου, θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα και να συζητήσουμε το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης και των νέων και της άμυνας που ανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μοντή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα επαναλάβω πολλά που είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον εισηγητή. όπως είπε ο κύριος Βιώτη και θα συμφωνήσω μαζί του, όταν κάνατε την πρόταση αναφερθήκατε στην ανάγκη ενίσχυσης ε, της προσπάθειας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης της προσπάθειας για τη σωστή εφαρμογή προγραμμάτων όπως το Horizon 2020 με την καλύτερη δυνατή χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Τώρα ειδικά για το ΕΦΣΥ και τη συνέχεια, νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει μια καλύτερη επεξεργασία της αρχής της ε, προσθετικότητας και τι ακριβώς έχουμε πετύχει στον τομέα αυτό μέσω του ΕΦΣΙ. Στα σημεία τώρα που έθεσαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι για το τομέα της ασφάλειας και άμυνας ε, κατανοώ ε, την λογική πίσω από αυτό αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν επιπλέον πόροι. Θα πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις εάν πράγματι θέλουν να τονώσουν την έρευνα στον τομέα αυτό. Και τέλος, όπως φαντάζεστε και εσείς, η συζήτηση για το Brexit, τους ιδίους πόρους κτλ είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ, συνάδελφοι, έκανα ό,τι μπορούσα πέρυσι για να παραμείνει η Ένωση στην Ένωση. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό θα ήταν για τη χώρα μου το καλύτερο στο μέλλον. Ίσως να παρατηρήσατε ότι <laughs> εγώ δεν ε, μπόρεσα τη θέση μου να την ε, κάνω να περάσει αλλά για το 18 η χώρα μου θα είναι μέλος και θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις τις δημοσιονομικές τις οποίες έχει. Αλλά αναγνωρίζω ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει ε, απομάκρυνση από τη λυγική του, της δίκαιης επιστροφής, του just retour. Λοιπόν, να τιμήσω την προσπάθεια που κάνατε, αλλά αν η Ευρώπη μιλούσε πιο ξεκάθαρα και στους Ευρωπαίους και τους Βρετανούς, θα μπορούσε κανείς να τεκμηριώσει την παραμονή στην Ένωση με καλύτερο τρόπο. Η κυρία Τομά. Η κυρία Τομά η οποία δεν είναι απελπισμένη αλλά λυπάται που η Ιταλική κυβέρνηση δεν ε, ήρε την επιφύλαξή της αυτό το οποίο με κάνει να λυπάμαι, λέει η κυρία Τωμά, είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι και αυτός ε, στο ύψος των περιστάσεων και το είπαν πολλοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μουρεσάν, με τον οποίο σε κάποιους τομείς συμφωνούμε, σε κάποιες προτεραιότητες συμφωνούμε. Όπως είπε και ο Σκιώδης μας, έχουμε και κάποια θέματα τα οποία συζητάμε ακόμα για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Να ξεκινήσω τώρα με μία απλή παρατήρηση πριν επανέλθω στη συνολική εικόνα τη δημοσιονομική. Η παρατήρηση αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι μια παρατήρηση κριτική στο σημείο 3 του εγγράφου. Ε, χρησιμοποιείται νομίζω μια επικίνδυνη διατύπωση. Λέτε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, μόνον αυτές μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Αυτό είναι ιδεολογικό περισσότερο το θέμα. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Θεωρώ όμως ότι είναι επικίνδυνη διότι δικαιολογεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης ε, την αντικατάσταση των επιδοτήσεων από τα χρηματοδοτικά μέσα. Ε, η λογική είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο τα χρηματοπιστωτικά μέσα και να μην υπάρχουν επιδοτήσεις καθόλου. Αυτό είναι σε αντίθεση και με το σημείο 11, όπου επιμένεται στην σημασία που έχουν οι πολιτικές συνοχή. Το ένα με το άλλο δεν είναι συμβατά. Τώρα θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις προτεραιότητες. Θα ήθελα να πω ότι η κύριε Φερνάντες για πρώτη φορά ίσως δεν συμμερίζομαι όλες σας τις προτεραιότητες. Καταρχάς, όπως είπατε, έχουμε έναν μικρούτσικο προϋπολογισμό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να γίνουν ε, κάποιες διαιτησίες. Οι διαιτησίες αυτές μπορεί να γίνουν και εδώ θα γίνει μια κάποια συζήτηση θα πρέπει να γίνουν ε, σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό τα ερωτηματικά εδώ είναι ανοιχτά. Εγώ θέτω τα ερωτηματικά και εγώ με τη σειρά μου χωρίς όμως να δίνω απαντήσεις. Κύριε Φερνάντες, αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια επιλογή, μια διαιτησία ανάμεσα σε διαφορετικές ανάγκες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν μειώσεις και αφαιρέσεις, οπότε και αυτό έρχεται και στον τομέα της άμυνας, όπως είπε και ο κύριος Γκέγερ και όπως είπε ο κύριος Ντανανό, δεν θα πρέπει να κάνουμε μεγάλους, μεγάλα, λέμε μεγάλα λόγια στον τομέα της άμυνας και να έχουμε έναν πολύ μικρό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι της άλλης θίγει άλλες δημοσιονομικές προτεραιότητες. Αυτό ισχύει κάθε φορά. Κάθε φορά μετά μεγάλα λόγια και ε, δυστυχώς λίγα χρήματα. Νομίζω ότι το είπανε πολλοί συνάδελφοι για το θέμα της άμυνας είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση και ίσως κύριε Πρόεδρε θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια συζήτηση και με την αρμόδια υποεπιτροπή του Κοινοβουλίου γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνειδητοποιούν σε καμία περίπτωση τις δημοσιονομικές συνέπειες των προτάσεών τους. Τελειώνοντας, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ κάτι το διφορούμενο στα πλαίσια των κατευθυντηρίων, στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της μετανάστευσης, ειδικά στον τομέα της μετανάστευσης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η ανθρωπιστική πολιτική ε, δεν υπογραμμίζεται όσο πρέπει. Δεν αναφερόμαστε στο Συριακό σαν παράδειγμα άμεσα και ίσως απαιτείται στο συγκεκριμένο σημείο μια προσπάθεια αναδιατύπωσης. Ευχαριστώ κύριε Τωμά, ο κύριος Μάγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισήγητη για την έκθεση του. Συμφωνώ με όλα, σχεδόν με όλα. Και στη τελική ανάλυση πιστεύω ότι η έκθεση θα είναι θετική. Θεωρητικά έχουμε πολύ καλά μέσα και εργαλεία στη διάθεσή μας. Αλλά αυτό που λείπει θεωρώ προσωπικά είναι ε, το βήμα της πρακτικής εφαρμογής. Και εδώ νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις χάνουμε το ρου της σκέψης μας. Χθες ε, είχαμε ε, αντιπροσώπους του Ταμείου Επενδύσεων του ΕΦΣΥ της Τράπεζας Επενδύσεων μας μίλησαν για παράδειγμα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων ενός δις ε, ύψους τα έξοδα και τα πάνε. Σε το ΕΦΣΥ μπορούν να το, να το, να το χρηματοδοτήσει. 95% προέρχεται από τα κρατη χρηματοδότηση και 5% από το ΕΦΣΥ. Και ο παράγοντας συντελεστής μόχλευσης είναι 19 φορές. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε όμως καλύτερα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Είναι καλό εργαλείο το ΕΦΣΥ σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι όμως σωστό να αφαιρούνται πόροι από την συνοχή και να προορίζονται και να διοχετεύονται σε αυτά τα προγράμματα. Επίσης αναφέρθηκαν και κάποιες ελλείψεις για την υλοποίηση. Το 2015 συζητήσαμε και αναφέραμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αναλύσεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν πληρώνει στην ώρα της τους λογαριασμούς της και έτσι προφανώς προκύπτουν καθυστερήσεις οι οποίες πλήττουν τους δημάρχους των μικρών του πόλεων. Τους αφήνουν νους και χωρίς χρήματα. Και προκαλούν όλα αυτά προφανώς αγανάκτηση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σχετικές αναλύσεις και να δούμε τι προγράμματα προωθούμε. Δεν έχουμε λάβει τέτοιες αναλύσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τώρα. Εμείς τα γράφουμε και τα λέμε, αλλά δεν υλοποιούνται. Η κυρία Τωμά ανέφερε τον τομέα της άμυνας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που δήλωσε. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να προβούν σε αγορά εξοπλισμού από κοινό. Και αν αυτό λειτουργούσε, θα μπορούσαμε κάθε χρόνο να απελευθερώνουμε πάρα πολλά χρήματα για τον τομέα της άμυνας. Έχουμε λοιπόν καλές ιδέες, αλλά πρέπει επιτέλους να υλοποιηθούν κιόλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μούρεσάρ, να πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η έκθεση και αυτά τα οποία είπατε για τις προτεραιότητες ε, σήμερα το πρωί ήταν πολύ καλά τεκμηριωμένα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ελάχιστες παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς αναφερθήκατε και εσείς στην ε, πολιτική συνοχή και αναφέρθηκε και ο κύριος Μούρεσαν στην πολιτική συνοχή. Πιστεύω ότι πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα και πρέπει να παραμείνει ως προτεραιότητα. Και γιατί αναφέρομαι στην πολιτική συνοχή τώρα. Διότι ανησυχώ για τα όσα είπε η κυρία Μέρκελ για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε με την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ελπίζω πραγματικά να μην είναι ε, αυτή η ε, δυσάρεστη συνταγή που συζητήσαμε και πριν από κάποια χρόνια ότι οι πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες ε, θα αναπτυχθούν ε, ταχύτερα και αυτές που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες δεν θα ακολουθήσουν. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συνταγή, χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία. η εμπορική και οικονομική συνεργασία λειτουργεί καλύτερα σε χώρες που όντως έχουν περίπου την ίδια οικονομική ανάπτυξη και έχουμε αρκετές χώρες ε, στις οποίες ε, το επίπεδο του ΑΕΠ είναι κάτω από το μέσο όρο και αν αυτές είναι οι δύο ταχύτητες τότε πρέπει να επιταχύνουμε αυτές τις χώρες στις οποίες η οικονομική ανάπτυξη είναι κάτω από το μέσο όρο. Και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό επιχείρημα η δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς με τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής. Κύριε Πρόεδρε, εσείς αναφερθήκατε στο Εράσμους. Το Erasmus Plus, ε, κατά την άποψή μου, είναι μια πολύ επιτυχημένη υπόθεση. Ε, φέτος ε, γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την έναρξη του Εράσμους. Είναι χρονιά επαιτίων, όχι μόνο τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα 30 χρόνια του Εράσμους. Ήδη 9 εκατομμύρια άνθρωποι ε, έχουν ε, ε, χρησιμοποιήσει το Εράσμους και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε αυξήσει και τους πόρους γιατί και πάλι θα αποτελέσει πολύ σημαντική όθηση για την ευρωπαϊκή οικονομία. Άκουσα επίσης για 6% διοικητικών δαπανών. Ε, και κάποιος είπε ότι είναι πολύ χαμηλός αριθμός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλό το ποσό και πρέπει να μειώσουμε τις διοικητικές δαπάνες, διότι Εγώ βλέπω μισθούς, ε, κοινωνικά επιδόματα, ε, δημοσίων υπαλλήλων και τον τρόπο με τον οποίο τα ξοδεύουμε. Πιστεύω ότι έχουμε περιθώρια και αν μειώσουμε τις δαπάνες αυτές, ο λαός ε, θα μας ευγνωμονεί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια με πολύ καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Merci. La parole est à Patricia Patricia Ευχαριστώ πολύ. το κύριο Μουρεσάν για την εξαιρετική έκθεση ε, η οποία είναι προσεχμένη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια όπως πάντα. Στον προπολογισμό του 2018 προσπαθούμε να επιτύχουμε στόχους όπως η αλληλεγγύη, η μετανάστευση, ανάπτυξη, θέση εργασίας, πολιτική συνεχής, ε, αλλαγή του κλίματος ε, και εράσμους. Στόχοι τους οποίους επικροτώ. Θεωρώ όμως ότι ξεχάσαμε την ευελιξία κάπου στον προπολογισμό. Το 2018 η ευελιξία του προπολογισμού θα είναι επαρκής ή αυτός ο προϋπολογισμός ε, θα πρέπει να καταρτιστεί με τρόπο ώστε να λάβουμε υπόψη και απρόβλεπτα, όπως για παράδειγμα ασφάλεια, άμυνα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές νέες ροές μεταναστών και προσφύγων, υπάρχουν αρκετές εγγύησεις για αυτά τα πρόβλεπτα. Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω αφορά τα αποτελέσματα. Είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτό το οποίο μας φέρνει τελικά ο προπολογισμός. Όλες οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται και μονογραφούνται είναι απαραίτητες, ε, διότι πρέπει να υπάρχει σαφής έλεγχος. Οποιοδήποτε λανθασμένο έργο αποτελεί ζημία για άλλον τομέα σε οικονομικό επίπεδο. Ε, πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού και γιατί ο προπολογισμό ε, είναι αρκετά περιορισμένος. Τρίτον, κατά την άποψή μου, Ε, πολύ σημαντικό είναι το θέμα των ιδίων πόρων. Η ομάδα Μόντι δημοσίευσε μία έκθεση για τους ίδιους πόρους όπως γνωρίζουμε. Τα επόμενα βήματα στο τομέα αυτό ε, μπορεί να είναι και πάρα πολύ αργά λόγω και της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό φυσικά με ανησυχεί. Και επίσης, πώς να αντιμετωπίσουμε τα κενά τα οποία θα προκύψουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα 16 περίπου δις ε, ευρώ τα οποία πληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο ετησίως στον προπολογισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση ο κύριος Όλμπριχτ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να ολοκληρώσουμε, εγώ θα είμαι λίγο πιο επικριτικός προς τον συνάδελφο, επειδή είμαι και από την ίδια πολιτική οικογένεια και μπορούμε να διαβάσουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε είτε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάποιον άνθρωπο μέσο άνθρωπο που δεν ξέρει τι συμβαίνει στον προπολογισμό και τα πράγματα είναι γενικά και κάνουμε τα συνήθη. Διότι ε, είμαστε στην έκτη χρονιά των δημοσιονομικών ε, προοπτικών. Δεν είμαστε στην πρώτη χρονιά, είμαστε στην έκτη. Ή μπορούμε να τα συζητήσουμε ω άνθρωποι του προπολογισμού, να καταλάβουμε λοιπόν τι υφέρπει και να δούμε ότι αυτή είναι στην πραγματικότητα συζήτηση για τον προπολογισμό εκβαθέων. Εγώ λοιπόν δεν κάνω μια ανάγνωση ω ε, γενική δήλωση για να είμαστε είμαστε καλύτεροι, πιο ανεπτυγμένοι κλπ. Αλλά ω τι θα θέλαμε να ζητήσουμε στου επόμενου μήνε. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Και γιατί αυτό. Πρώτον, διότι η αναθεώρηση δεν ήταν μια συμβολική διαδικασία, ήταν αναθεώρηση η οποία ήταν έτοιμα προς το Συμβούλιο ότι χρειαζόμαστε ένα πιο ευέλικτο προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή για το 2018 χρειαζόμαστε ευελιξία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευελιξία. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το 18. Αν οι Ιταλοί δεν αλλάξουν άποψη και αν δεν αλλάξουμε άποψη εμείς αν δεν αλλάξουν οι Ιταλοί, θα έχουμε πάλι μια κατάσταση χωρίς ευελιξία και τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα γίνει με τις προτεραιότητε αν δεν έχουμε ευελιξία. Ο κύριος Μουρεσάν λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε τις προτεραιότητε, αλλά να ξέρουμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεύτερον, αυτό είναι το πρόβλημα, για παράδειγμα, της πολιτικής συνεχής. Αναφέρεται η περιφερειακή πολιτική στο κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι προτεραιότητα. Ακούστηκε αυτό προηγουμένως. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο προπολογισμό του 17 έχει μείωση στη συνοχή κατά 25% για το 17 στις πληρωμές. Το 2018 λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση στις πληρωμές. Το ερώτημα είναι ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού θα παραμείνει το 2018 για τη συνοχή όταν γίνεται τόσο σημαντικό άλμα σε αυτές τις πληρωμές. Αν κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο με το 2017, τότε θα έχουμε αμέσως καθυστέρηση. Ε, και η στέρηση πληρωμών. Εάν τα συγκρίνουμε ε, σε σχέση με το 2017, μπορεί να σωθούμε. Το θέμα είναι αν το Συμβούλιο θα είναι διατεθειμένο να διπλασιάσει το κονδύλιο για, τον, για τη συνοχή το 2018. Διότι αν διπλασιάσουν το κονδύλιο για τη ε, συνοχή το 2018, τι θα μειώσουν. Το συμπέρασμα είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερε πληρωμέ. Χρειαζόμαστε περισσότερε πληρωμέ στον προπολογισμό. Αλλιώ θα βρεθούμε παγιδευμένοι. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μούρεσαν που είπε ότι μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το κείμενο λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτές είναι οι προτεραιότητές μας, αυτά θα ζητήσουμε και μην περιμένετε από εμά να ε, παρατηθούμε κάποιων ετοιμάτων. Εάν δεν παρατηθούμε όμως θα πρέπει να ε, δώσουμε όθηση στον προπολογισμό του 18. Είναι η πέμπτη χρονιά αυτή και είμαστε και ένα χρόνιο πριν ε, από το Brexit και επιπτόντως δεν είναι 16 τα δις ε, μετά τους, ε, την αποχώρηση των Βρετανών, θα είναι 5 δις. Αν δούμε τις επιστροφές, τις πληρωμές και τις δαπάνες κλπ, στην ουσία ο λογαριασμός βγαίνει 5 δις. Μην υπερβάλλουμε και μόνοι μας. το θέμα είναι κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν αυτό το, τα 5 δις μετά την αποχώρησή τους. Συνοψίζω. Θεωρώ ότι το κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα ε, σαφές πολιτικό μήνυμα, δεν είναι πολύ σαφές για τους ανθρώπους που δεν ε, καταλαβαίνουν, γιατί νομίζουν ότι επαναλαμβάνουμε τα τετριμένα. Πρέπει όμω να κάνουμε και μια δεύτερη ανάγνωση και να τα δούμε πολύ πρακτικά και πολύ συγκεκριμένα. Γιατί αλλιώς, ε, όπω είπε και ο κύριος ε, Μάνκα χθε, ε, συζητούσαμε για το ΕΦΣΙ. Κάποιο από του εμπειρογνώμενε είπε ότι αν δεν τα δίνετε στη συνοχή να τα βάλετε στο Ταμείο στρατηγική ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων. Ε, Κάποιο είπε πάρτε τα από τη συνοχή και δάστε τα εκεί γιατί είναι πιο αποτελεσματικά. δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Αν αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε με τις δικές μας ε, προτεραιότητες, γιατί η συνοχή είναι επιμερισμένη διαχείριση και επομένω είναι και δική μας αρμοδιότητα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και η δομή του προπολογισμού του 18 είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι πολύ πιο δύσκολη από το 17. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι είναι μια δύσκολη χρονιά για τις κυβερνήσεις. Μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις στους δημόσιους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνουν τις πληρωμές. Και βλέπουμε στο τέλος του χρόνου ότι υπήρχαν επιστροφές προς τις κυβερνήσεις. Καλό ήταν αυτό. Λειτουργούσε η Ευρώπη και η συνεισφορά ε, του προϋπολογισμού βέβαια δεν ήταν ε, ιδιαίτερα σημαντική. Και γι' αυτό ακριβώς ε, το 2018 ήταν κάτι το, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τα πράγματα και θα έχουμε μια έκρηξη στις πληρωμές. Όλα αυτά βέβαια είναι εντελώς αμφισβητήσιμα. Για μα, όμως ε, η αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ε, τουλάχιστον αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ε, απαιτεί ομοφωνία. Αυτό είναι το βέβαιο. Όμως για την ε, συνδιαλλαγή στον προπολογισμό δεν χρειαζόμαστε ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Ίσως λοιπόν θα πρέπει ε, επειδή δεν θα υπάρξει αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου στη συνδιαλλαγή να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις της αναθεώρησης ε, που είχαμε συζητήσει όταν την ονειρευόμασταν και να προσπαθήσουμε να τα διαπραγματευτούμε αυτά μέσω μιας ε, ειδική πλειοψηφία. Και εδώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μόρισαν για να μας κάνει παρατηρήσεις για να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρα και εν συντομία από δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια που έκαναν. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμα τα σχόλια αυτά και αυτή είναι η δική μου η άποψη και πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας από τώρα μάλιστα από την φάση των τροπολογιών προς την έκθεση αυτή και που θα προσθέσουν θεωρώ σημαντικά στοιχεία. Και όπως είπατε και είπε και ο κύριος ε, Ολμπριχ και η κυρία Τωμά και εσείς πρόεδρε θα πρέπει να έχουμε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Το πώς θα αποφασιστεί λοιπόν ο προπολογισμό στο επόμενο έτος και πώς θα υλοποιηθεί. Και στο πνεύμα αυτό λοιπόν αναφέραμε τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην αποχώρηση του, της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα όσα έγιναν στην ομάδα υψηλού επίπεδου και την αναθεώρηση του τρέχοντος πολιτισμού δημοσίκου πλαισίου. Θα συμμετέχουμε λοιπόν στις ε, συνδιαλλαγές, θα έχουμε πάντα υπόψη μας το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε, μεταξύ άλλων και την αναθεώρηση του τρέχοντος ε, του δημοσιονομικού πλαισίου. Και ασφαλώς θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες συνέπειες των προπολογισμών για του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τον Brexit, φυσικά ο αντικτύπος ε, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι μηδαμινός, ε, πολύ μικρός, 0,5. 0,1% γιατί το Brexit δεν θα γίνει του χρόνου προφανώς. Μέχρι να σημειωθεί το Brexit λοιπόν και να υλοποιηθεί θα είναι πλήρες μέλος η, Ευρωπα... Βρετανία και απόλυτα δεσμευμένη στη συνεργασία μαζί μας. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική τώρα συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στον προπολογισμό, θα έχω να πω το εξής. θα πρέπει να είμαστε ε, σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και τις δεσμεύσεις μας, αλλά να είμαστε και να έχουμε υπόψη μας και τις ε, επιπτώσεις των προπολογισμών. Για του χρόνο, λοιπόν θα είναι μη η επιδρασή. Αυτά, συνάδελφοι, και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία, στις τροπολογίες που θα λάβω την επόμενη τρίτη στις 6 το απόγευμα λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και μετά στις 6 Μαρτίου θα το συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστώ και προβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Γενικό Εισηγητή. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήπως έχουν κάποια παρατηρήση να μοιραστούν μαζί μας. Μήπως κάποιους νέους πόλους που θα μας επιτρέπαν να επεκτείνουμε κάποιο φάκελο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, η οποία κατέδειξε θεωρώ ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύγκληση σε ό,τι αφορά τους στόχους και σύγκληση και με τις προτεραιότητες που έχει ορίσει έως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες προτεραιότητε, επιτρέψτε μου ίσως για κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση προκειμένου να μην υπάρχουν και παρανοήσεις για την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων δεν φρενάρει ουσιαστικά την πληρωμή των ε, λογαριασμών. Και ο κύριος Μάνκα ε, είπε ότι δεν έχουν γίνει αναλύσεις. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι μετά από εντολή του Κοινοβουλίου εφαρμόσαμε ένα σχέδιο πληρωμών το οποίο μας ε, επέτρεψε να ρυθμίσουμε την κατάσταση έως τώρα έχουν πληρωθεί λοιπόν τα τιμολόγια και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε διαφορά της πιστώση. Το 2018, ωστόσο, θα πρέπει να επιταχυνθούν τα προγράμματα συνοχής και πάλι. Αυτό αποτελεί μια μεταβλητή που καθορίζει το συνολικό επίπεδο πληρωμών και προφανώς θα υπάρξει αύξηση. Αυτό αναμένουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τους νέους αυτούς τους ρυθμούς. Θα αναλάβει λοιπόν τις ευθύνε της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για τα έργα του 2018. Μία τελευταία παρατηρήση. Για τα καταπιστευματικά ταμεία, τα trust fund για το οποίο επικρατεί κάποιος σκεπτικισμός από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αναφέρθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας υπενθυμίσω ότι έχει δεσμευτεί για τον προπολογισμό του 2017 ο Επίτροπος Oettinger τίμησε τη δεσμεύση αυτή που είχε αναλάβει με επιστολή προς εσάς κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στα συμβούλια των Trust Funds και Επίσης, ό,τι αφορά την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου για την υλοποίηση και την εκτέλεση των Trust funds. και θα ήθελα να έχουμε ανοιχτό πνεύμα σε ό,τι αφορά τα trust funds, γιατί τα trust Funds αποτελούν μια απάντηση σε συγκεκριμένες ε, προκλήσεις και επιτρέπουν ε, τη χρήση των πόρων και τον καλύτερο συντονισμό με τις δράσεις ε, των κρατών μελών στα θέματα για τα οποία προορίζονται. Αυτές οι παρατηρήσεις εκ μέρους μας λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Και χαιρετίζουμε και πάλι το έργο του εισηγητή καθώς και τη συζήτηση που έγινε. Ευχαριστούμε. Αν μπορέσετε να μας στέλνετε ένα σύντομο ε, σημείωμα για την χρηματοοικονομική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ε, αυτή την διευκόλυνση του προπολογισμού που βρισκόμαστε εμείς, αυτό το budgetary facility και τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Οι δεσμεύσει είναι 3 δι ή 6 δι ε, και ποιο είναι ο τρόπος ε, χρηματοδότησης. Ωραία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων λοιπόν. Ήταν διαφωτιστική η παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μόρεσάν. Περνάμε τώρα σε μία ανακοίνωση του Γενικού Εισηγητή μας για το 2016 για την αλληλεγγύη. Βλέπουμε ότι η αλληλεγγύη με το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ε, πραγματικά ζωηρή, κάτι το οποίο θα παρηγορήσει την κυρία Μούντι. Κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η αλληλεγγύη πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Η πρότασή μου στοχεύει σε μια επιτάχυνση της υιοθέτησης της συγκεκριμένης πρότασης. Καλούμε ε, ε, το Συμβούλιο να ακολουθήσει και αυτό μια εξίσου ταχεία ε, διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας ε, την αποστολή αυτή. Θα πρέπει τα ποσά τα οποία έχουν ε, καθοριστεί να μπορέσουν να φτάσουν στους δικαιούχους στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πορτογαλία, ιδιαίτερα στην αυτόνομη περιοχή ε, της Μαντέιρα. Το ποσό είναι 63 εκατομμύρια ευρώ. Ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο και 4 περίπου 3,9 εκατομμύρια για την Πορτογαλία. Ε, δεν έχει ζητήσει προκαταβολή το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περίπτωση όμως της Κύπρου και της Πορτογαλίας ε, ξέρετε ότι υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές. Στην Κύπρο επίσης υπάρχει και το θέμα της ξηρασίας και εξ αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έκθεση θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνει δεκτή έτσι ώστε ε, τα ποσά τα οποία είναι προκαθορισμένα να φτάσουν στις τρεις αυτές χώρες ε, το ταχύτερο δυνατόν και επαναλαμβάνω στην Πορτογαλία, στην περιοχή την αυτόνομη της Μαδέιρα. Ο προϋπολογισμός λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία ακόμη φορά δείχνει ότι είναι ένας προϋπολογισμός αλληλεγγύης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μετά από φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς οι φυσικές αυτές καταστροφές εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ σοβαρές και προέρχονται από τις κλιματολογικές αλλαγές. Θέλει κάποιος το λόγο για την έκθεση Φερνάντες, όχι. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιος. Ε, υπάρχει συνένεση πλήρης. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν πριν από τις 2 Μαρτίου στη μία το μεσημέρι. Αλλά θα πρέπει όπως είπαμε να πάμε αρκετά γρήγορα και γι' αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν θα ψηφίσει την πρόταση στις 30 Μαρτίου αλλά στις 20-21 Μαρτίου. Αυτό θα έχει σαν επιπλέον πλεονέκτημα να είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι του ΕΛΚ γιατί στις 30 Μαρτίου θα βρίσκονται όλοι στην Ίσο Μάλτα για το κογκρέσο του κόμματος. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στις 26 ή στις 27 Απριλίου. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Γκέιερ. Ο κύριος Γκάγερ θα μας μιλήσει για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαρίθμου 1. Κύριε Γκάγερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, στην προκειμένη περίπτωση κινούμαστε όπως και μέσα στη μεταφορά που μίλησαμε προηγουμένω. Η συνέπεια για το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι μια αλλαγή του που θα κινητοποιήσει ένα ποσό για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και Αλληλεγγύη, το οποίο μόλι ανέφερε ο κ. Φερνάνδε, μην τα επαναλαμβάνω όλα αυτά. Υπάρχει ένα μικρό λάθο ό,τι αφορά τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ θεωρούμε ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ε, δεν στέκουν τα ποσά των ε, προκαταβολών που δόθηκαν στα κρατημέλη και αυτό το επικρίνω και στο κείμενό μου. Η Μάλταζικη Προεδρία δεσμεύτηκε ότι θα διορθώσει το σφάλμα αυτό. Θα λάβουμε δηλαδή τα σωστά στοιχεία και κατά τη λήψη των αποφάσεων θα διαγράψουμε την προκειμένη παράγραφο γιατί πλέον δεν θα έχει α, ε, ουσία. Τεχνικό πρόβλημα. Που ωστόσο πρέπει να επιτυπωθεί. Θα πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν έχω και τίποτα άλλο να σας πω οι προθεσμίες είναι οι ίδιες με αυτές του Χωσέ Μάριο, γιατί επί της ουσίας ε, σύνδεονται τα θέματα. Ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή και δεν βλέπω να υπάρχουν και σχόλια. Μιλάμε για την υλοποίηση της έκτασης την οποία μας παρουσίασε ο Χωσέ Μανουέλ. Οι ημερομηνίε λοιπόν 2 Μαρτίου στις 1 το μεσημέρι για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στην ημερομηνία που ανέφερα προηγουμένως για την έκθεση του Χωσέ Μανουέλ και το ίδιο και για την Ολομέλεια στο Στρασβούργο τον Απρίλιο. Η κυρία Χολμάιερ θα έρθει. καθυστερούμε λίγο το θέμα της και θα δώσουμε και πάλι το λόγο στο Γενικό Εισηγητή, τον κύριο Γκάιερ, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης ε, Επαγγελματικής Κατάρτισης, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Κύριε Γκάιερ. Πρόεδρε, ε, αν μου επιτρέπετε θα πρότεινα τα τρία επόμενα σημεία στην ημερήσια διαταξή να τα πραγματευτούμε από κοινού, το 10, 11 και 12 δηλαδή γιατί συνδέονται και πάρα πολύ μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αντίρρηση, λέει ο πρόεδρο. Μιλάμε για την τροποποίηση των ε, βασικών κανονισμών ε, των υπηρεσιών αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν να κάνουν με την απασχόληση σε μεγάλο βαθμό. Το Σεντεφόπ είναι η υπηρεσία που ασχολείται με την επαγγελματική κατάσταση. Η Eurofund ε, εξετάζει τους όρους εργασίας και η όσα επίσης συγκαταλέγεται στο ίδιο πακέτο σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου πρόκειται για μια διαδικασία η οποία αφορά αυτές τις συνδεόμενες υπηρεσίες και την τροποποίηση του βασικού κανονισμού. Θα πρότεινα λοιπόν στην Επιτροπή Οι τροπολογίες που θα γίνουν για την τροποποίηση των κανονισμών να είναι και για τις τρεις υπηρεσίες. Και η βασική γραμμή είναι ότι όπου υπάρχει δυνατότητα συνεργασία μεταξύ των τριών οργανισμών, θα πρέπει να ενισχύονται και σε αυτές συγκαταλέγεται και ο σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για το ποιο οργανισμό είναι υπεύθυνο και αρμόδιο Γιατί, για να μην υπάρχουν άλλες επικαλύψεις και να τα κάνουμε όλα δύο φορέ. Σε περίπτωση που εργάζονται οι παραπάνω οργανισμό για κάποιο σημείο. Έκανα λοιπόν κάποιε προτάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο των ε, Υπηρεσιών προτείνω να συμπεριλαμβάνονται και μέλη από τα Διοικητικά Συμβούλια των άλλων υπηρεσιών. Να υπάρχει διάλογος για το ποια εργασία μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά σε ποιον οργανισμό. και για την καλύτερη δικτύωση των οργανισμών με τα άλλα όργανα. Σημαντικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει η... ο ρόλος παροχής υπηρεσιών των οργανισμών αυτών. Τροπολογίες μέχρι την άλλη εβδομάδα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και στις 20-21 Μαρτίου θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τις εκτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για τις ε, επεξηγήσεις αυτές, οι οποίες ε, έχουν να κάνουν με την τροποποίηση των βασικών κανονισμών και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Όλμπριχτ ζήτησε καταρχάς το λόγο. Θα ήθελα να μεταφέρω τις απόψεις του σκιώδους εισήγητού μας του κυρίου Σάβαρμα συμφωνεί με τις ε, προτάσεις ε, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αποφυγή επικαλύψεων ανάμεσα στις τρεις αυτές ε, εξωτερικές υπηρεσίες. Ζητά συγγνώμη γιατί δεν είναι εδώ ο ίδιος. Αυτά. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος άλλος, ο κύριος Κάμελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γκάιερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οργανωθούμε καλύτερα, να δημιουργηθούν συνεργασίες προκειμένου να μην υπάρχει έλλειψη συντονισμού να μην υπάρχει παράλληλη δράση. Άρα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Αλλά πιστεύω ότι οι τρεις αυτοί οι τομείς οι οποίοι δείξατε και οι οποίοι συζητιούνται είναι οι κατεξοχήν τομείς στους οποίους ισχύει ε, η αρχή της επικουρικότητας. Ε, εντάξει, τους έχουμε αυτούς τους οργανισμούς. Τι κάνουν όμως ουσιαστικά και όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, σημαντικές διαφορές συγγνώμη, μεταξύ των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος πηγαίνει διακοπές σε κάποιο άλλο κράτος μέλων, διαπιστώνει, για παράδειγμα, πόσο διαφέρουν ε, τα πράγματα μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Ερωτώ, λοιπόν, και διερωτώ μου, πραγματικά σκοπός μας είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ορίσουμε προδιαγραφές οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες σε κάποια κράτη στην παρούσα φάση. Δεν μπορούν πολύ απλά να τα πληρώσουν. Μήπως θα έχει πιο πολύ νόημα να κάνουμε λίγο πιο πίσω και να προβαίνουμε σε πιο λίγες συστάσεις, λίγες συστάσεις οι οποίες θα ήταν πιο ρεαλιστικές σε ό,τι αφορά την υλοποίησή τους. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν χώρε που θα δυσκολεύονταν να τι υλοποιήσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε με μεγάλη, με πολύ αυστηρό και κριτική διάθεση το τι μπορεί να παραλυφθεί και τι όχι. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς ζητάει το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες από τις ε, τροπολογίες και να ζητήσω από τον εισηγητή να τις λάβει υπόψη του όσο μπορεί. Παρά το γεγονός ότι επικροτούμε τις προτάσεις και την ιδέα και το στόχο για καλύτερη συνεργασία και αποτελεσματικότητα, έχω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, συνέπεια με τους κείμενους κανόνες. Στην ε, κοινή προσέγγιση των αποκεντρωμένων οργανισμών που αποφασίστηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτοί που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο των Οργανισμών ε, αναφέρονται ως εκπρόσωποι κρατών μελών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου ενδείκνυται. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια αναφορά σε ε, συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπου των θεσμικών οργάνων. Επιφυστώ λοιπόν την προσοχή σας σε αυτή την τροπολογία που ε, θα ε, επιτρέπει να έχουμε εκπροσώπους από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Δεύτερον, ένα σημείο για την τροπολογία υπερθμών 6. Αναφέρεται την ε, ε, πράξη χρηματοδότησης για τα κέντρα μετάφρασης που λέει ότι τα κέντρα μετάφρασης θα πρέπει να παρέχει ε, μετάφραση σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες και οργανισμούς. Στην τροποποίηση λέγεται τώρα ότι η ε, μετάφραση θα πρέπει να παρέχεται από το κέντρο μετάφρασης ή άλλες υπηρεσίες παροχής μεταφράσεων. Εδώ μπορεί να υπονομεύσουμε το ρόλο του κέντρου μετάφρασης, ε, το οποίο στην ε, πραγματικότητα έχει αρμοδιότητα να παρέχει αυτές τις μεταφραστικές υπηρεσίες στους άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες. Και τέλος θα ήθελα... Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία υπαριθμών 8 Υπάρχει μια φράση που λέει ότι προς αυτό το σκοπό η υπηρεσία θα παρέχει ε, συμβουλές και υπηρεσίες και προτείνεται ο όρος services, υπηρεσίες, να αντικατασταθεί από τον όρο ανάλυση. Αυτός είναι στην ουσία ο ρόλος των τριών υπηρεσιών, αλλά για την περίπτωση της ΕΝΤΕΦΟΠ Μπορεί να υπάρχει κάποιος περιορισμός, διότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, παρέχει και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση του Europass ε, και ε, διαχειρίζεται και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες για την απόφαση για το Europass, καθώς επίσης διαχειρίζεται και το σύνολο δεδομένων του λεγόμενου European Skill Panorama. Δεν ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, ε, να χαθούν φυσικά αυτές οι αρμοδιότητες του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ε, δεν φαντάζομαι ότι ήταν αυτός ο σκοπός της τροπολογίας, αλλά να φροντίσετε ίσως να έχετε μία διατύπωση που θα επιτρέψει στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ να συνεχίσει με, αυτές, με αυτά τα καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρέζα. Κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις ε, παρεμβάσεις σας. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κόλμελ. Να σας πω το εξή. Ε, σωστά οι παρατηρήσεις σα, ωστόσο δεν επηρεάζουν τις αρμοδιότητες σε καμία περίπτωση των συγκεκριμένων οργανισμών. Τι κάνει η Eurofund. Μας παρέχει, για παράδειγμα, και αυτό αποτελεί ένα από, τα σημαντικά, από τις σημαντικές του ε, οργανισμού. Μία επισκόπηση του τι γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι τόσο ετερογενή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει κάποια συγκρισιμότητα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη μέθοδο συλλογή στοιχείων, αλλά, για παράδειγμα, με το ποιον τρόπο συλλέγονται τα δεδομένα στα κρατημέλη μελη Και αν θέλουμε να έχουμε ε, μια επισκόπηση της πολιτικής, της κοινωνικής κατάστασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίληψη για το τι γίνεται, προκειμένου να υπάρχει και πολιτική να ξέρουμε τι γίνεται και από πολιτικής άποψη. Και είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να απασχολούμε 28 διαφορετικού ε, παράγοντες στα κράτη-μέλη, οι οποίοι στη συνέχεια θα συλλέγουν στοιχεία τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να διαμορφώνονται με κάποιο συγκρίσιμο τρόπο. Και έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένας ενιαίος οργανισμός και αυτό είναι πιο φτηνό από το να υπάρχουν 28 αντίστοιχες εθνικές αρχές οι οποίες να εξοπλίζονται. Το ίδιο ισχύει και με το Συντεφόπ. Και εδώ δεν ε, θεωρούμε ότι υπάρχει το θέμα που αναφέρατε. Αν θέλουμε οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πραγματικά την δυνατότητα μετακίνηση και να είναι πραγματικά ελεύθεροι και να βρουν μια θέση απασχόληση σε κάποια άλλη χώρα, χρειάζεται μια κεντρική τέτοια ευρωπαϊκή αρχή που θα το εγγυάται αυτό. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, είναι πιο λογικό να γίνεται από μια κεντρική υπηρεσία παρά από 28 εθνικές ε, υπηρεσίες. Άρα εδώ πέρα η επικουρικότητα δεν θεωρώ ότι είναι πραγματικά σχετική. Προς τον κύριο Πρέντα να πω το εξή. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να χάσει στο στο ΣΥΝΤΕΦΟΠ ξαφνικά επειδή δεν έχουμε κάνει τις ε, σωστές ε, νομικές διατυπώσεις για την τροπολογία 6 ε, για τα κέντρα μετάφρασης. Να σας πω ότι αυτό αποτελεί μία μόνιμη πηγή διαμάχης μεταξύ μου ως ε, εισηγητή και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί το κέντρο μετάφρασης ε, δεν είναι πλέον σε θέση, λόγω των αλλαγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ανταπεξέλθει στην ταχύτητα των μεταφράσεων. Και πολύ απλά έτσι έχει κατάσταση. και αυτό πάντα εκφράζεται στα διάφορα έγγραφα στις απαλλαγέ και ούτω καθεξή, στο θέμα τη μείωση του προσωπικού. Σε κάποιες ε, περιπτώσεις οδηγεί σε απόλυτη απόδοση και αυτό έγινε στο κέντρο μετάφραση. Δεν μπορώ να πω ότι υπολειτουργούν. Θα ήταν υπερβολικό αυτό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ ε, είναι συχνό το φαινόμενο να περιμένουν ε, υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα διάφοροι οργανισμοί για μεταφράσει. Και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό κλάδο, ξέρετε ότι ο χρόνο όντω είναι χρήμα. Ή ενδεχομένω να οδηγεί σε κριτική αυτό, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλο το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένουν ε, οι υπηρεσίε. Αυτό δεν το λέω για να τονίσω την σημασία του κέντρου μετάφρασης, αλλά για να έχουν τις ε, υπηρεσίες, οι οργανισμοί αυτοί, τις υπηρεσίες μετάφρασης στη διάθεσή του. Γιατί πολύ απλά, αν δεν προλαβαίνουν να γίνουν μεταφράσεις, καθυστερεί όλη η εργασία. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική που ακολουθούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η εναλλακτική θα ήταν να επεκτείνουμε και να πάρουμε πιο πολλού μεταφραστέ. Αλλά δεν μπορώ να το προτείνω αυτό στην παρούσα φάση. Πρέπει να το κοιτάξουμε το 2008. Η κοινή προσέγγιση, έχετε δίκιο, δεν μιλάει για τα διοικητικά συμβούλια κτλ. Αλλά θεωρούμε ότι σκοπός ε, δεν είναι να διαταράξουμε τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων. Μπορούμε, για παράδειγμα, να προτείνουμε ρόλο παρατηρητή στα διοικητικά συμβούλια. Αλλά θεωρώ ότι όταν μια οργάνωση έχει ένα παρόμοιο και συναφές πεδίο εργασίας με κάποια άλλη οργάνωση και θα μπορούσε να ενημερώνεται εγκαίρως για τον τρόπο λειτουργίας μιας άλλης οργάνωσης, ε, αυτό θα ήταν ωφέλιμο. για να ξέρει ποιε είναι και οι προθέσεις των άλλων οργανώσεων πρωτού. Ε, συγχωρέστε με αν ε, θεωρείτε ότι είμαι επιθετικός, αλλά αν υπάρχει χώρος για 28 εκπροσώπους των κρατών μελών στα διοικητικά συμβούλια, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι σε κάποιε περιπτώσει ε, είναι πιο πολύ στο Διοικητικό Συμβούλιο παρά οι εργαζόμενοι και πάλι της, ε, του οργανισμού. Υπερβάλλω λίγο, αλλά όχι πολύ. Ε, θεωρώ ότι είναι προφανέ το πώ μπορούμε να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψει στι περιπτώσει αυτέ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό και έτσι μπορούμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, στις 20 Μαρτίου να ψηφίσουμε. Ε, υπάρχει, υπάρχει χρόνο, υπάρχει ε, προθεσμία για τις 16 Φεβρουαρίου 11 η ώρα για τις τροπολογίες και από εκεί και πέρα η συζήτηση θα γίνει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις μας. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω το Γενικό Εισηγητή αν είχαμε κάποιες εξελίξεις ε, με την Ελλάδα για το θέμα των, ε, της μετεγκατάστασης των οργανισμών. Υπήρξε κάποια κίνηση από αυτό ή να το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Η Μόνικα Χολμάιερ εδώ για να συζητήσουμε την πολιτική για τα κτίρια και ίσως να ψηφίσουμε κιόλα. Κυρίως για το Κοινό Κέντρο Έρευνας και το σχέδιο στην Ίσπρα, στην Ιταλία. Κυρία Χολμάιερ, θέλετε να παρέμβετε, παρακαλώ. Θα σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το Joint Research Center 102 με έδρα στην Ίσπρα, μια κοινή ερευνητική α, υπηρεσία. Με μια σειρά την οποία παρακολούθησα την προηγούμενη θητεία, πρέπει να σας πω ότι η Ίσπρα έχει ένα πανάρχαιο κτίριο χτίστηκε κάπου μεταξύ της δεκαετίας του 50 και του 80 και φαίνεται. και στη συνέχεια ε, προστίθενταν συνέχεια μικρά κτίρια κοντά στο αρχικό. Και πλέον ε, έχουμε 11 κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται Και μιλάμε και για κτίρια τα οποία χρησιμοποιούν και κάνουν έρευνα ε, την ενεργή κτλ. Κτίρια 44-37 χρονών και δεν έχει νόημα να διατηρηθούν όλα αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα κτίριο 10.500 τετραγωνικών μέτρων. Καθαρή επιφάνεια όμως, με εργαστήρια δηλαδή και γραφεία 6.400 τετραγωνικών μέτρων. Ανά άτομο έχουμε περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα μέγιστη χωρητικότητα 345 άτομα, ενώ τώρα έχουμε 315 άτομα. Και από τον προπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν 3,9 εκατομμύρια ευρώ. 19% μόνο. Δεν χρειάζεται ξένη χρηματοδότηση. Γιατί έχουν τα έσοδα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται με την πάρδο των χρόνων. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τα assigned revenues ε, μειώθηκαν τόσο πολύ μεταξύ του 2013 και 2014, γιατί είχαμε 13,6 εκατομμύρια. Από το 2014 είμαστε στα 5,6 και πλέον να υπάρχει μια μικρή άνοδος, κάτι πάνω από 9 εκατομμύρια. Γιατί τόσο μεγάλη αλλαγή μεταξύ του του προγράμματος ε, πλαίσιο, του 7ου προγράμματος πλαισίου και του ορίζοντα 2020. Θα ήταν ενδιαφέρον από πλευρά προπολογισμού να το ξέρουμε αυτό, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα όλων αυτών πληρώνεται ακριβώς από αυτά τα εκχωρημένα έσοδα. Θεωρητικά λοιπόν ε, είναι σημαντικό να μπορούν να τα παρανούν οι πόροι αυτοί και για την έρευνα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το τι πετυχαίνουμε με τα, με τις εκορυμένες, ε, τα έσοδα. Γιατί διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για χώρες όπως το Ισραήλ, η Βοσνία Σεχοβίνη, το Ισραήλ, η Φαράω, η Μακεδονία, όλες αυτές είναι συνδεδεμένες χώρες. Και σε τελική ανάλυση αυτά τα εκπορημένα έσοδα χρησιμοποιούνται ως ε, βοηθητικό εργαλείο για να μην έχουμε ξένες, ε, ξένο κόστος. Και να μπορέσουμε να βοηθηθούμε σε τομείς όπου τα κρατημέλη θα είχαν καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την πληρωμή για τα κτίρια. Και έτσι λοιπόν θα ήταν δύσκολο να γίνουν τέτοιες, ε, να υπάρχουν τέτοιες και το, το καταφέρνουμε λοιπόν αυτό μόνο με τα εγχωρημένα έσοδα. Και έτσι λοιπόν έχουμε πλέον ε, αρκετά τέτοια έσοδα ειδικού προορισμού. Και αυτό μειώνει το συνολικό κόστος, γιατί μιλάμε για ένα κεντρικό κόστος και έτσι θα είχαμε 747.000 ως έξοδα. Περιλαμβάνονται λοιπόν διάφορες δυνατότητες σε διάφορα τα κτίρια. Θα πρέπει να πούμε ότι από πλευρά ε, αποδοτικότητας ε, χρειαζόμαστε μείωση του κόστους, ε, σημειώνεται μάλλον μείωση του κόστους κατά 60% λειτουργικού κόστους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι πολύ απλά βγάζει νόημα. Και η κεντρική διαμόρφωση στα πλαίσια του ΙΣΠΡΑ θα γίνει και στο μέλλον, αλλά το θέμα είναι τα ενεργά απορρίμματα από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που καταφέραμε, μεταξύ άλλων και με πίεση της Επιτικής μας Επιτροπής, είναι ενδιαφέρον ότι η δική μας Επιτροπή είναι αυτή που πίεσε. Πριν από πολλά χρόνια, ξέρετε, ξεκινήσαμε να θέτουμε το ερώτημα τι είδους ραδιενεργά απόβλητα υπάρχουν και έκτοτε καταγράφονται όλα. Μεταφέρονται σε μια διάμεση αποθήκη. Έχουμε πλέον επίγνωση του τι ακριβώς περιλαμβάνεται, πόσο ραδιενεργό είναι. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η κεντρική πλέον καταχώρηση και που η Ιταλική κυβέρνηση πιέζει για μια λύση καθοριστική. Γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχει ένας ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο και μετά να παραδοχιόνται τα υλικά εκεί πέρα. Όχι, θέλουμε να ξέρουμε να υπάρχει σωστό έλεγχο σωστή υποπτία σε όλη την ε, φάση. Και αυτό το αναφέρω ω θετικό στοιχείο στην παρούσα φάση, γιατί πριν από κάποια χρόνια δεν ίσχυε. Αυτό δεν είχε βέβαια να κάνει τίποτα με το κτίριο και με την οικοδόμηση των κτιρίων, αλλά ήθελα να πω ποια είναι η θετική επίδραση τη επιτροπή μα. Έτσι, επιτέλους, με την πίεσή μας ε, είναι μεγαλύτερη και πιο η αντιμετώπιση από την ΙΣΠΡΑ και στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλο το κείμενο. Ευχαριστώ κυρια Χόλμαγερ. Θέσατε το ερώτημα και για τους πόρους που έχουν διατεθεί. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να δώσει απάντηση, ο κύριος Πρέζα ίσως. οι συνάδελφοι του Κοινού Κέντρου Έρευνας να δώσουν τις απαντήσεις αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρισήμιση λιγότερο για το Κοινό Κέντρο Έρευνας. In addition, during the years 2014... σε σχέση με το 2014, για την περίοδο μάλλον, 14-16, η Ελβετία δεν πήρε μέρος στο Horizon 2020, μόνο σε τμήματα που δεν αφορούν στον προϋπολογισμό του Κοινού Κέντρου Έρευνας. Concerning the commissioning, we have characterized and identified all the waste we have in ISPRA, and we have moved all this to... Νομίζω ότι για τα απόβληπα της Ίσκρα έχουμε σε ενδιάμεση ε, αποθήκευση και περιμένουμε τη συνεννόηση με τις Ιταλικές αρχές για τη διάθεσή τους. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες, με τον σωστό ελπίζω τρόπο. Κοιτάξτε, οι, διατεθέντες περνάνε από 3% σε, από 30% συγγνώμη, σε 25%. 14 εκατομμύρια το χρόνο, λέει ο εκπρόσωπος του Κοινού Κέντρου, αλλά από το 14 αυτό έγινε ε, 5 εκατομμύρια μόνο, οπότε έχουμε ένα κενό για το 15 και το 17 μείον 8 εκατομμύρια και εδώ ελείπουν για το 17 10 εκατομμύρια λόγω της μη συμμετοχής της Ομοσπονδίας της Ελβετικής. Μπορώ να σας διαθέσω τα αριθμητικά στοιχεία των 7,7 δις και στη συνέχεια πήγε στα 13,6 εκατομμύρια και στον ορίζοντα 2006 πήγε στο 5,3 και τώρα σιγά σιγά αυξάνεται το ποσοστό στον 9,9 αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι η συμμετοχή στον τομέα αυτό έχει περιοριστεί. Γι' αυτό λοιπόν το επισημαίνουμε ότι στον ορίζοντα 2020 και στα προγράμματα και εντομίας θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ως Επιτροπή Προϋπολογισμού για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα γιατί με κάθε ε, λεπτό και ευρώ που λείπει, έχουμε και λιγότερα έσοδα ειδικού προορισμού και μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλο και λιγότερα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι άλλε χώρε. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σαφέ και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιδείξουμε την απαραίτητη προσοχή. Merci pour ε, cette... Ε, Ευχαριστούμε που κρούεται τον κόδον του κινδύνου. Όσον αφορά το θέμα της προετοιμασίας του προπολογισμού, της κατάρτισης του προπολογισμού, αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, αυτό είναι στα έσοδα ή είναι στη μείωση των δαπανών στον προπολογισμό. Είναι μάλλον ε, η δεύτερη περίπτωση, δηλαδή είναι στις δαπάνες ε, και Εκεί αναφέρονται τα ποσά τα οποία προβλέπονται για αυτά τα έσοδα ειδικού προορισμού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη ε, για να υπάρχει, αν θέλετε, φρέσκο χρήμα στον προπολογισμό. Δεν είναι ανομαλία του προπολογισμού αυτού, διότι κανονικά αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται στα έσοδα και στις δαπάνες ε, θα έπρεπε να αναφέρεται το σύνολο του ποσού. είναι στη στήλη των δαπανών ακριβώς για να αιτιολογήσει το αίτημα ε, του, ε, της έγκρισης της πίστοσης. Διότι ξέρετε ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το ύψος των δαπανών είναι αυτό το οποίο καθορίζει τα ε, ύψος των εσόδων και τη συνεισφοράς που ζητάτε από τα κράτη-μέλη ε, και από εκεί και πέρα στα έσοδα λαμβάνονται υπόψη άλλα έσοδα αλλά αυτά αφορούν κάποιες δαπάνες και δεν αναγράφονται ως έσοδα. Ο κανόνας αυτός είναι γενικός. Τα έσοδα είναι αυτά τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό και ήδη οι πόροι χρησιμοποιούνται για ε, την πληρωμή του συνόλου των εξόδων ε, χωρίς να αφορούν κάποια συγκεκριμένη δαπάνη κάθε φορά. Ναι, μεν, αλλά ήσασταν εκεί όταν, ε, παρόν όταν έγινε η συζήτηση για το σχέδιο προπολογισμού του 18 και τους προσανατολισμού που συζήτησε ο, ειδικός, ο, Γενικός Συγητής είπε ότι αυτός ο τρόπος είναι ε, αδύνατο να τον ε, αντιληφθεί ένας απλός πολίτης. Και νομίζω ότι αυτό το σύστημα των εσόδων ειδικού προϋπολογισμού καταδεικνύει ακριβώς ότι ε, μειώνουμε στην πράξη τον αριθμό των δαπανών που εμφανίζονται στο προϋπολογισμό θα πρέπει να εξηγήσουμε και τι τύπο ε, εσόδων ειδικού προορισμού έχουμε. Για παράδειγμα, αν συμμετέχουν χώρε όπω η Ελβετία ή μια τρίτη χώρα σε κάποια προγράμματα, στην πραγματικότητα αυτά τα έσοδα ειδικού προορισμού είναι ένας τρόπος ε, πληρωμής ε, για τη χώρα αυτή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν προβλέπονται στην αρχική νομική βάση που καλύπτει τις ε, χώρες μέλη, αλλά εδώ έχουμε συμμετοχή και τρίτων χωρών που συμμετέχουν και αυτά με τη δική τους την ποσόστοση. Για λόγους διαφάνειας λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχουν ε, παρεκκλήσεις από τους στόχους των δαπανών. Από την άλλη υπάρχει το άλλο παράδειγμα της διευκόλυνσης για την Τουρκία που αναφέρατε προηγουμένως. Εκεί έχουμε... Ε, διμερή συμμετοχή από πλευράς κρατών μελών για την πολιτική αυτή και προβλέπουν ε, ποσό βοήθεια το οποίο υπερβαίνει αυτό το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους και τα έσοδα του προϋπολογισμού. Ε, όσον αφορά τη διαφάνεια λοιπόν και τις ε, αιτιολογήσεις νομίζω ότι αυτά ε, έχουν μια σωστή λογική στον προϋπολογισμό. Ε, δεν ξέρω, οι εμπειρογνώμονες μπορεί να το καταλάβουν, οι απλοί πολίτες δεν ξέρω. Πρόεδρε, να πω ότι κάπου δεν διαφωνώ, αν μου επιτρέπετε. Γιατί, αν μια χώρα προδεσμεύεται για να συμμετέχει με ένα ποσό σε ένα πρόγραμμα, το κάνουν αυτό φυσικά με τη γνώση ότι χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά και για τα κτίρια και τα λειτουργικά έξοδα. Υπάρχει διαφάνεια και διατηρούνται τα στοιχεία αυτά για πενταετή περίοδο. Άρα θεωρώ ότι ε, από πλευρά ε, διαμόρφωση έχει νόημα να υπάρχουν έσοδα ειδικού προορισμού. Ε, ε βγάζει νόημα τώρα το γεγονό ότι δεν έχουν πάντα και τα κρατημέλη, εδώ θα συμφωνήσω. Ναι, υπενθυμίζω απλώ μία αρχή ε, καθολικότητα του προπολογισμού. Όλε οι δαπάνε ε, χρηματοδοτούνται από το σύνολο των εσόδων. Θα έχουμε βέβαια ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε δέχομαι την πρακτική γιατί είναι αυτή η οποία προβλέπεται και από τον κανονισμό αλλά αν θέλουμε ο προϋπολογισμός ε, να γίνεται εύληπτος από τους πολίτες ε, και συμμετέχει και μια άλλη χώρα, παραδείγματος χάρη Ελβετία, καλό είναι να υπάρχει μια σαφήνεια για την ισορροπία στον προπολογισμό. Περνάμε σε ένα ε, σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να ε, ψηφίσουμε. Παρακαλώ τις συναδέλφους να μείνουν στην αίθουσα για να υπάρχει απαρτία. Ε, και η απαρτία είναι σχεδόν στο κόκκινο. Σας παρακαλώ λοιπόν μείνετε στις θέσεις σας. Κυρία Χολμάιερ, πιστεύετε ότι πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Ε, συγγνώμη, κάτι μου είπε ο συνάδελφο και ήθελα να το απαντήσω και. Ναι. Σα Ζητούν ε, λοιπόν την προσοχή σας από άλλο. Θέλετε να ψηφίσουμε? Πολύ ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ε, διάταση του της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν στη χρηματοδότηση αυτή. Μας παρουσίασε η κυρία Χόλμαρη τις λεπτομέρειες. Ποιοι είναι λοιπόν υπέρ. Ο Γενικός Εισηγητής για το 2018, κύριε Μούρεσαν, Υπέρ ή κατά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι είμαι υπέρ. Πολύ ωραία. Ομόφωνα λοιπόν. Ακολουθούμε την πρόταση της κυρίας Χολμάιερ. Κυρία Χολμάιερ, έχετε το λόγο τώρα για τη Frontex. Ένα δεύτερο έργο το οποίο μας απέστα, αλλά και το ακόμα δεν θα το ψηφίσουμε σήμερα. Μία ενημέρωση η Frontex ε, μας ε, έστειλε τα μελλοντικά στοιχεία με αρκετά διάφανη τρόπο. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ε. Και αυτά θέλουν να μας τα πούν σε μια κανονική ενημέρωση και να ψηφίσουν αυτά στη συνέχεια. Μιλάμε για την έδρα στην Βαρσοβία. Όλοι ξέρουμε ότι η Frontex θα έχει πολύ περισσότερο προσωπικό πλέον και στην Βασοβία και η κατάσταση λοιπόν έχει ως τώρα, ως εξή. Από τους 14 ε, ορόφους ε, η Frontex έχει 9. 14.600 τετραγωνικά μέτρα, 14 συνεδριακές αίθουσες, υπάρχει μία καντίνα στον 14ο όροφο, Το πρόβλημα είναι ότι δεν του στάνουν οι όροφοι. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεταβατική κατάσταση. Μέχρι ότου οικοδομηθεί ένα καινούριο, εντελώ καινούριο κτίριο στην Πολωνία το 2022. Η BNP Paribas που έχει τον δεύτερο μέχρι και τον πέμπτο όροφο στο κτίριο αυτό και αυτή προγραμματίζει νέα κτίρια. Θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι αυτή η εννέα όροφη είναι στο ιδιοκτήριο. Το μόνο που είναι πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα για την Frontex αυτό, είναι ότι έχουμε εκμίσθωση των κτηρίων αυτών μέχρι το 2024, ενώ εμεί θέλουμε να μετακομίσουμε το 2022. Τι θα γίνει λοιπόν τα δύο επιπλέον αυτά χρόνια. Θα ήθελα να έχω λοιπόν πιο πολλές πληροφορίες. Αν μετακομίσουμε το 2022, τι θα κάνουμε, θα πληρώνουμε μέχρι το 2024 ε, τα χρήματα για την εκμίσθωση των ορόφων αυτών. Αυτό φυσικά δεν μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά ενδεχομένω να μην μπορέσουμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση μίσθωσης και να χρειαστεί να πληρώσουμε πρόστιμα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση, να κοιτάξουμε τι λεπτομέρειε και να πληροφορηθούμε για τι λεπτομέρειε. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει σήμερα. Απλά ήθελα να προειδοποιήσω τη Frontex ότι θα θέλαμε πιο πολλέ πληροφορίε για το θέμα αυτό. Και ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρέ διαπραγματεύσει. Γιατί αυτά που προβλέπονται ω πρόστιμα είναι λίγο προβληματικά. Και να δούμε κατά πόσο η Πολωνία όντως ε, θα έχει ολοκληρώσει μέχρι το 2022 το κτίριο. Μάλλον θα διαθέσει το οικόπεδο για να χτίσει το κτίριο όπως έχει υποσχεθεί. Αυτό θα πρέπει ενδεχομένω να το κοιτάξουμε στις διευκρινήσεις. Όπως σας είπα, σήμερα είναι μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε πριν την ψηφοφορία σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δηλαδή συμβόλαιο και ανάλογα με τις συνθήκες που θα έχει πετύχει η Frontex. Το ίδιο αποφάσισε και το Συμβούλιο και θεώρησε ότι αυτή η πρώτη ενημέρωση ήταν ε, συμβατή με τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Frontex ε, χρειάζεται κάτι καλύτερο, κάτι πιο σημαντικό και φυσικά θα χρειαστεί χρόνος για την κατάλληλη υποδοχή στη Βασεβία. Εν τω μεταξύ όμως οι πολωνικές αρχές υπέγραψαν την συμφωνία για την έδρα για να μπορέσει η Frontex να υποδεχθεί και νέους συνεργάτες ε, που μέχρι τώρα ε, δεν ήταν τόσο εύκολο να έρθουν διότι ε, έλειπε μια διάταξη που δεν επέτρεπε να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να υπάρχουν διάφορα ωφέλη που προσφέρονται στους εκπακτηριστέντες. Υπήρξε όμως επίσημη δέσμευση των πολωνικών αρχών που επιτέλους υπέγραψαν τη συμφωνία για την έδρα της Frontex στη Βερσονία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Δεν έχει υπεγραφεί, λέει η κυρία Χολμάιερ. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιε δυσκολίες για την πολωνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διάθεση από την πολωνική κυβέρνηση αυτού του κοπέδου 20 δισεκατομμυρίων σκοπεύουν να το κάνουν, αλλά ως τώρα δεν με έχουν ενημερώσει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο συγκεκριμένα, δηλαδή να έχουν πραγματικά δώσει το οικόπεδο αυτό. Ο κ. Λετζέρε μου αναφέρει ότι είναι ακόμα σε συζητήσεις, οι οποίες πάνε καλά, δεν λέμε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ληφθεί η οριστική απόφαση. Ναι, για το οικόπεδο. Για το οικόπεδο. Ναι, αλλά όταν μιλάω για τη συμφωνία, για την έντρα, μιλάω για τη συγκεκριμένο καθεστώς που θα έχουν οι πράκτορες που θα είναι στη Βαρσοβία. Για παράδειγμα για τα προνόμια που θα έχουν τα φορολογικά, για τα σχολεία των παιδιών τους, οτιδήποτε θα μπορούσε να ανακόψει τη μετακόμιση των, της, της στην ε, Βαρσοβία. Άλλο για το οικόπεδο. Ναι, και εδώ όμως υπάρχουν κάποια έκρεμη ζητήματα, γιατί η κυβέρνηση ε, δεν είναι τόσο δυναμική όσο ήταν ε, τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Θα τα ξανασυζητήσουμε γιατί ούτω ή άλλω η απόφαση αναβάλλεται. Ε, δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Ε, θα ακούσουμε την κυρία Γκαρδία Θαμπάλ τώρα να μας διευκρινίσει τα της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων και τις ε, ε, δραστηριότητές της, κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ε, προηγούμενη φορά η παρουσίαση ήταν ιδιαίτερως διαφωτιστική. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεισέφερε σε επενδύσεις στην Κίνα, σε επενδύσεις στο Χονγκ Κόνγκ, για παράδειγμα. Καλή και άγια η διάθεση να δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάζεται πιστώσεις ε, για να ε, καλύψει δάνεια τα οποία εν μέρη χρηματοδοτούνται από την Κίνα και ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει στην Κίνα, το βρίσκω πραγματικά εκπληκτικό. Είναι επενδύσει που συνεισφέρουν στη βελτίωση του κλίματο, μου είπατε. Τότε φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα βοηθά και τι επιχειρήσει ε, τη Ευρωπαϊκή να επενδύσουν στην Κίνα. Η απάντηση ήταν ότι όχι. Ε, τέλος πάντων αυτό πρέπει να συζητηθεί και θα ήθελα να ξέρω λίγο και τον δικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύριε Αγκαρδία Θαμπάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, για το, τις χώρες τις οποίες επενδύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ποιες είναι οι πολιτικές ε, και οι στόχοι της, ε, σε αυτές τις επενδύσεις ε, είναι τμήμα αυτών ε, των οποίων συζητούμε εδώ σε αυτή την έκθεση για την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τις προάλλες, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, ήδη έγινε μια συζήτηση για τις γενικές γραμμές ε, και άκουσα και τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Έθεσα και μια σειρά από ερωτήματα και βάσει και τη συζήτηση που έγινε και βεβαίως και βάσει και των προτάσεών μου, ε, ε, πρότεινα και μια σειρά από τροπολογίε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. 35 τροπολογίε, 34 για την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων και μόνο μία για το Ταμείο Εγγυήσεων. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειε για κάθε μία, αλλά ε, στην ουσία... αφορούν πέντε θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι τα ποσά τα οποία διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορέσει να επενδύσει σε ε, επενδύσεις στις χώρες αυτές. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ή άλλως αύξανε τα ανώτατα όρια για τις επενδύσεις αυτές, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πάμε ε, έτη περαιτέρω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι με ένα μικρό ποσό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μπορούμε να αυξήσουμε κατά πολύ τα δάνεια τα οποία ε, μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτές τις χώρες. Και προτείνω να γίνει αυτή η άξιση κυρίως ε, διότι τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουν σχέση και με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπήρξαν δύο πολύ σημαντικές κρίσεις, τις οποίες βιώσαμε στην περίγυρό μας. Ε, μία στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρειάστηκε να ενισχύσει και να προκαταβάλει όλες τις επενδύσεις στο πρώτο τμήμα του πολιτικού σχεδίου και φυσικά η προσφυγική κρίση η οποία δεν έχει μόνο συνέπειες εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ε, σε όλες τις χώρες ε, της γείτονο περιοχής. Επομένως, ε, πιστεύω ότι με αυτή τη μικρή αύξηση στον προπολογισμό μπορούμε να αυξήσουμε κατά πολλού τις επενδύσεις σε αυτές τις γειτονικέ χώρες. Δεύτερον, η δεύτερη ενότητα τροπολογιών ε, έχει σχέση με το νέο στόχο που προτείνεται στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί μία έκφραση η οποία λέει να αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε τις βασικές βαθιές αιτίες της μετανάστευσης. Είναι μία φράση την οποία ακούμε σαν το Ευαγγέλιο εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν είναι σαφές το τι υπάρχει πίσω από αυτήν την άποψη ε, που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της μετανάστευσης. Γιατί αν δούμε τους τρεις στόχους που περιλαμβάνονται στην πρόταση της τράπεζας, δηλαδή ανάπτυξη του τοπικού ιδιωτικού τομέα, βοήθεια προς τις μικρομεσαίες, ε, βοήθεια προς τις υποδομές κοινωνικές και οικονομικές, μεταφορές, ε, ενέργεια, εκπαίδευση υγεία και υγιεινή, καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών, όλα αυτά είναι μορφές καταπολέμησης των αιτιών. Και γι' αυτό ο τέταρτος στόχος θα πρέπει να διατυπωθεί, να γίνει κάπως πιο συγκεκριμένος, να έχει δηλαδή σχέση ε, με την φροντίδα όλων των μεταναστών και ιδιαίτερα των προσφύγων ε, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες υποδέχονται ε, τους ε, μετανάστες, τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα τις χώρες οι οποίες λειτουργούν σαν σημείο περάσματος των προσφύγων. Ήδη λοιπόν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές αυτό έχουν σαν στόχο να καταπολεμούν την ε, μετανάστευση μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών αυτών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν ίσως κατάλληλο να τροποποιήσουμε αν θέλετε την ονοματολογία του τέταρτου αυτού στόχου γιατί ήδη περιλαμβάνονται οι προηγούμενοι στόχοι. Η πρόταση αυτή ξέρω ότι θα προκαλέσει ίσως αρκετές συζητήσεις, αλλά η συζήτηση θα είναι ε, ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τις εξωτερικές εντολές της ε, τράπεζας, αλλά και για τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες ε, στα πλαίσια του Ταμείου Επενδύσεων. Επίσης ε, σε σχέση και με την πολιτική των φύλων, την διάσταση του φίλου, αυτό δεν άπτεται μόνο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επενδύσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έννοια του φύλου, τη διάσταση του φύλου. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται και στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούμε. Ένα τέταρτο μπλοκ, μια τέταρτη ομάδα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, προσοχή και υπογράμμιση της σημασίας των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον τύπο των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτούνται και κατά πόσον αυτές θα επηρεάζουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το τελευταίο θέμα είναι το θέμα της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, φορολογικών παραδείσων, φορολογικής διαφθοράς κτλ. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται προγράμματα ε, τα οποία να χρησιμοποιούν ενδιαμέσους οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε και να ενισχύσουμε και να αυξήσουμε τους ελέγχους μας και την πολιτική μας η οποία είναι κατά της φοροδιαφυγής και κατά α, της μη σωστής χρήσης των φορολογικών μέσων. Να πω λοιπόν τελειώνοντας ότι στην, για το Ταμείο Εγγυήσεων ζητείτε να υπάρξει μια μελέτη για την καταλληλότητα των νέων ποσοστών των εγγυήσεων, για τον τρόπο χρησιμοποίησης του Ταμείου αυτού και για τον τρόπο εφαρμογής του Ταμείου αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλιά σας και τις τροπολογίες σας και να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Ευχαριστώ κυρία Γουαρία Ζαβάλ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο, ο κύριος Μορεσάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρόταση την οποία έχει κάνει και για την προσπάθεια την οποία κάνει τους τελευταίες εβδομάδες. Και εμείς εξετάζουμε προσεκτικά τις προτάσεις για την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ακριβώς η βάση για να προχωρήσουμε. Πιστεύουμε ότι η εξωτερική εντολή θα πρέπει να καλυφθεί σε αυξημένο ποσοστό και πιστεύουμε ότι το επίπεδο το οποίο προτείνει η ίδια η τράπεζα είναι το κατάλληλο. Πιστεύουμε επίσης ότι η τράπεζα είναι σε καλή θέση ε, για να αξιολογήσει ακριβώς τις ανάγκες που έχει και τις ανάγκες αύξησης των δανείων προς ε, τρίτες χώρες, εκεί όπου είναι οι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την ουσία της πρότασης ότι το σύνολο να χαρακτηριστεί σε 38,5 δις. Τίθεται τώρα το θέμα πού θα πάνε τα χρήματα αυτά, σε ποιες χώρες και σε ποιες περιφέρειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξουμε κάποιες προτεραιότητες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα περιορισμένα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας στις περιοχές όπου οι επιπτώσεις των οικονομικών συνθήκων για την Ένωση και για το πληθυσμό της Ένωσης είναι ο πιο σημαντικός μέσω της σταθεροποίησης των τοπικών οικονομιών. Βλέποντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τις προτάσεις τις οποίες κάνει η συγγήτρια, ε, θα ήθελα να πω ότι εγώ προτιμώ τις προτάσεις της EIB που θεωρούν ότι ανάμεσα σε όλες τις περιφέρειες τα περισσότερα ποσά θα πάνε στη νότια γειτονία, 12,3 δις ευρώ, κάτι το οποίο είναι δικαιολογημένο λόγω της μεγάλης σημασίας την οποία έχει με η Μετσογειακή περιοχή για τα επόμενα χρόνια ε, στον τομέα της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφυγικών ρευμάτων από την Αφρική. Νομίζω ότι συμφωνούμε με την πρόταση ότι το ποσό αυτό είναι το κατάλληλο κατά τη, για την εντολή της CIB και δεν συμφωνούμε με την εισηγήτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθεί το ποσό αυτό κατά 1,3 δις επιπλέον. Συμφωνούμε επίσης με την εισηγήτρια για τους άλλους γεωγραφικούς τομείς, Ασία, Κεντρική Ασία, Νότια Αφρική. Ε, υπάρχουν κάποιες διαφορές όμως για τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Γειτονία. Ε, για την ανατολική γειτονία η τράπεζα ζητά περισσότερα χρήματα. Και βλέποντας την επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τις επιθέσεις εις βάρος της Ουκρανίας και το πολιτικό πλαίσιο έχουμε τρεις χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει μια στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία με εταιρικέ σχέσεις που είναι η στενότερη μορφή συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε με χώρες εκτός της Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την πρόταση της τράπεζας για αύξηση της εμπλοκής μας στην ανατολική γειτονία. Γνωρίζουμε ότι αν εμπλοκή ε, της τράπεζας συνεχιστεί, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, η οποία καταναλώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά αν θέλετε, αν συνεχιστεί λοιπόν στα επίπεδα τα οποία έχουν ε, επιβεβαιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, τα ποσά αυτά δεν θα αρκούν και γι' αυτό συμφωνούμε για μια ακόμη φορά με το αίτημα της τράπεζας να αυξηθούν τα ποσά για την Ανατολική Γειτονία. Και για τη Λατινική Αμερική ζητούνται περισσότερα χρήματα, σημαντικά περισσότερα, από 2,5 δις σε 3 ε, δις. Ε, είναι σημαντικό, θα το εκρίνουμε, αλλά δεν εγκρίνουμε την πρόταση της εισηγήτριας για μεγαλύτερη αύξηση αύξηση 20% για τη Λατινική Αμερική, 500 εκατομμύρια επιπλέον για μια περιοχή η οποία δεν είναι στην άμεση γειτονία μας με την οποία έχουμε όμως ε, σχέσεις αλλά έχουμε άμεσα θέματα ε, στη γειτονία μας και στο νότο και ανατολικά όπως το προτείνει η τράπεζα. Η αύξηση λοιπόν για τη Λατινική Αμερική πρέπει να γίνει όπως το λέει η IB αλλά όχι όπως λέει η Θα συμφωνήσω λοιπόν με τις προτάσεις της εισηγήτριας ε, για να αυξηθεί και η παρουσία γενικότερα της, ε, να αναγνωριστεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας όπως επίσης και να υπάρξει μια σωστή ε, αναγνώριση της σημασίας της, της προβληματικής του φύλου. Αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς όμως να επιβάλλονται επιπλέον βάρη διοικητικά στην τράπεζα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αρνητικές ε, επιπτώσεις. Αυτά τώρα για το Ταμείο Εγγυήσεων. Εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την άποψη της εισηγήτριας και αυτή είναι η άποψη και της Επιτροπής ότι μακροπρόθεσμα η χρήση των ποσών αυτών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος. Νομίζω ότι θα, η μετακίνηση ε, της διαχείρισης του Ταμείου θα κοστίσει 4 εκατομμύρια ε, εφάπαξ και από εκεί και πέρα 1 εκατομμύριο το χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένας καλός στόχος. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παρούσης εντολής. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο όφελος σε επίπεδο κόστους, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με τον εισηγητή τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, σαν μακροπρόθεσμη πρόπτικη, συμφωνώ με τον εισηγητή και την Επιτροπή. Αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για το σχέδιο αυτό και για τις ιδέες που μας παρουσίασε, με τις οποίες ε, πρέπει να σας πω ότι επί της αρχής σύμφωνα τις βρίσκω καλές. Θα ήθελα να τονίσω και άλλη μια πτυχή στη συζήτηση επιτρέψτε μου να κάνω μία αναδρομή στην ε, μεγάλη κρίση που ζήσαμε το 2007 και 2008. Στη Γερμανία, να σας πω ότι έχουμε 16 κρατήρια, ομόσπονδα, και κάθε ομόσπονδο κρατήριο κατά το παρελθόν είχε την αίσθηση ότι θα έπρεπε να συστήσει δική του κεντρική τράπεζα. Το κάναμε λοιπόν αυτό και ξεκινήσαμε δηλώνοντας ε, ότι, για παράδειγμα, η Βαντεμιτεμβέργη και η Κεντρική Τράπεζα προαγάγει τα δικά της έργα. Και σε κάποια φάση λοιπόν ξεκίνησαν να αναρωτιούνται γιατί να περιοριζόμαστε μόνο στη Βάντη Βιτεμβέργη, γιατί να ε, μην κάνουμε πολύ περισσότερα. Και έτσι άρχισαν να κάνουν διεθνώς ε, συναλλαγές τι σημαίνουν συναλλαγές, σημαίνουν και κίνδυνο και ρίσκο. Όλοι ελπίζουμε να μην α, ε, ε, εκπληρωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, αλλά κάποιοι εκπληρώνονται κιόλα. Και κάποιε λοιπόν πτώχευσαν. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το λέει και ο τίτλος της. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάθε συναλλαγή που εκτελείται συνεπάγεται και ένα ρίσκο. Αυτό να το αντιλαμβανόμαστε. Και κατά δεύτερον θα πρέπει να πληρώσουμε. Να προσέξουμε λοιπόν, να προσέξουμε προκειμένου να είναι Διαφανίσει οι δαπάνε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός σκιώδους προπολογισμού σε τέτοιες περιπτώσεις ε, που δεν προβάλλεται στον προπολογισμό. Αυτό ως σκέψη το καταθέτω. Είμαι βέβαιος ότι όταν δεν έχουμε πόρους στον προπολογισμό πρέπει κάπως να παρέχουμε την εγγύηση τα πρώτα χρόνια είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που δυστυχώς πρέπει να πληρώσουμε και το λογαριασμό. Να προσέχουμε λοιπόν και να φροντίσουμε να δώσουμε κάποια συγκεκριμένα σχόλια όσον αφορά την προσαρμογή αυτού του 9%. Καλύπτει αυτό του κινδύνους που αναλαμβάνουμε. Και για να μας δώσει κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, ε, αναφερόμαστε σε ρίζες ε, της μετανάστευσης, μήπως θα έπρεπε να αναφερόμαστε σε πηγές ε, μετανάστευσης, γιατί οι ρίζες φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τις πηγές. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες ο κύριος Μάρκος Πέρτ, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Τραπέζας Επενδύσεων την κυρία Καρδιά Θαμπάλ για την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία κατά την άποψή μου η οποία θα βοηθήσει την τράπεζα να ε, επιτύχει τις ε, πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, είτε για δραστηριότητές μας στη Λατινική Αμερική. Ε, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Η δήλωσή σας, η πρότασή σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το πιο βασικό και αποτελεσματικό μέσο είναι αυτή η πολιτική και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε πολύ μεγάλη επιρροή. Ε, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόταση που αφορά ε, της, ε, το warehousing γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την πρωτοβουλία για τη μετανάστευση, τη λεγόμενη πρωτοβουλία οικονομικής ε, προσαρμογής που είναι ζωτική σημασία για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Να καθησυχάσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κινείται προ αυξημένη διαφάνεια και είμαστε στη διάθεσή σα για να τα συζητήσουμε αυτά περαιτέρω. Τέλος, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να προλάβουμε την... Ε, ε, διεύρυνση των μέσων ε, ε, προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Μέσο Ρευστότητας είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει και πρέπει να διατηρηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα της εξωτερικής μας πολιτικής ε, πάντα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μήπως θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι. Θα ήθελα να πω κάτι. Καταρχάς ε, χαιρόμαστε για την πρόταση στην αύξηση ε, της εγγύησης, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 35 εκατομμύρια σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά το warehousing, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση, δεν υπάρχει κάποια πρόταση για την τροποποίηση της ε, ε, νομοθεσίας για να το διευκολύνουμε αυτό ε, που περιλαμβάνει η πρόταση του Συμβουλίου. Απλώς να πούμε ότι εμείς ήδη Έχουμε αυτή την πρωτοβουλία της οικονομικής προσαρμογής, έχουμε γκρίνει ήδη προγράμματα και ίσως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εγκρίνουμε προγράμματα που θα μπορούσαν να επωφεληθούν αυτές τις εγγύησεις αν υπάρχει κάποια εξασφάλιση ότι θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί και αναδρομικά η δυνατότητα αυτή για να μετριάσουμε τους κινδύνους που συνοδεύουν αυτά τα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα πρόγραμμα στο Λίβανο ε, για το Συμβούλιο του Μαρτίου αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επωφεληθούμε και της ε, ε, αναδρομικής εφαρμογής αυτής της εγγύησης, αλλιώς θα πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνούμε με την ανάγκη να ενισχύσουμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες ε, των ε, εκθέσεων ε, και της αξιολόγησης των έργων και υπάρχει και μία πρόταση αυτά τα φύλλα αποτελεσμάτων να δημοσιοποιούνται ανα έργο. Ε, αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι καλή ιδέα την οποία υποστηρίζουμε ε, και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τι επιρροή έχει το πρόγραμμα. Το θέμα είναι όμως ότι κάθε τέτοιο φύλλο είναι απλώς μία εκτίμηση όλων αυτών των οποίων περιλαμβάνονται σε ένα ε, πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και κάποια θέματα εμπιστευτικότητας, ε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται ότι το πρόγραμμα έχει τις ε, εξή αδυναμίες και προτείνονται κάποια πράγματα για να αντιμετωπιστούν, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε και κατάλληλη αξιολόγηση όλων αυτών. Όσον αφορά τις τροπολογίες ε, για ε, φορολογικές περιφέρειες που δεν ε, ε συμμορφούνται προς την νομοθεσία, ε, υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθούμε και στον τομέα αυτό. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία εδώ είναι να υπάρχει κάποια σαφήνεια περί του τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος, ε, υπάρχουν κάποιοι κατάλογοι που περιλαμβάνουν χώρες ε, που μπορεί να είναι και χώρες μελή ή χώρες όπως η Τουρκία και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως σας έλεγα, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει και σαφής ε, καθοδήγηση. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες που αφορούν τις ε, ε, πτυχές της ισότητας των φύλων. Ήδη έχουμε κάποιες πολιτικές επ' αυτών, όπου μπορούμε προσπαθούμε να αναφέρουμε και τα στοιχεία της ισότητας των φύλων και πρόσφατα εγκρίναμε και μια στρατηγική περισσότητας των φύλων που στόχο έχει να αντιμετωπίσει θέματα φύλου στις δραστηριότητές μας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Α, Συγγνώμη, συγγνώμη. Για τις ρίζες της μετανάστευσης, όπως ξέρετε, εμείς ως τράπεζα για τη μετανάστευση, όπως είπαμε και προηγουμένως, εμείς μπορούμε να δούμε κατά πόσον προσαρμόζονται οι χώρες φιλοξενίας και οι κοινότητες φιλοξενίας, ε, αλλά εκφύσεως ε, η τραπεζική εμπλοκή αφορά τις μακροπρόθεσμες πτυχές. Δεν είμαστε μάλλον εμείς σε θέση να απαντήσουμε σε ανθρωπιστικά ζητήματα, αλλά αν δείτε τα διάφορα προγράμματα ε, τα οποία υλοποιούμε σε αυτές τις περιοχές, μπορούμε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις σχετικές δομές και να υποστηρίξουμε και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα για να υποστηρίξουμε τη συνοχή. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις ρίζες της μετανάστευσης, αλλά και τις ε, ε, συγκεκριμένες ανάγκες ε, η φιλοξενίας, διέλευσης και λοιπά της κοινότητας των προσφύγων. Ο κύριος Ανζέλ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη φωνή μου. για την αύξηση του ανωτάτου ορίου. Σημειώνουμε την πρόταση της, της εισηγήτριας. Ξέρετε ότι υπάρχει μια κάποια αβεβαιότητα για τη δυνατότητα που έχουμε εμείς στα πλαίσια του παρόντος δημοσιονομικού πλαισίου να διασφαλίσουμε την άφηξη αυτή. Ιδιαίτερα μετά από τον Brexit, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε. Έχουμε πάνω από το κεφάλι μας ένα τεράστιο, ε, μια τεράστια σπάθη του δαμοκλέους δυστυχώς. και ιδιαίτερα για το τίτλο 4 δεν έχουμε κανένα περιθώριο σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα μπορέσει να διασφαλίσει ένα επίπεδο επέμβασης, αλλά έχουμε αμφιβολίες για την ε, δυνατότητα ε, του προϋπολογισμού να καλύψει ε, με τον τρόπο που το κάνει σήμερα την ανάγκη της τώρα για τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες. Ε, συμφωνούμε με την πρόταση του Κοινοβουλίου, η οποία συμπίπτει με τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συζητήσεις που έκανε. Μέχρι τώρα, όπως είπε ο συνάδελφος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μπει στον τομέα αυτό σε μια διαδικασία αλλαγής. Ήδη από πέρυσι υιοθετήσαμε ένα νέο έγγραφο για μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες που είναι θα έλεγα ένα πρώτο θετικό βήμα. Συνεπώς λοιπόν προσπαθούμε εμείς να διασφαλίσουμε με σωστό τρόπο τις ανάγκες μας για να μπορέσουμε ε, να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά ε, σε θέματα όπως η φοροδιαφυγή, και φοροαποφυγή κτλ. Τώρα, για την έδρα είναι σε ένα κράτος μέλος, στο Λουξεμβούργο. Απαντά στην ερώτηση του Προέδρου εκπρόσωπος τράπεζας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ότι αν πράγματι είμαστε σκληρότεροι ε, σε σχέση με τη χρήση των δικαιοδοσιών offshore, το κάνουμε αυτό για να προστατεύσουμε ε, τα συμφέροντα των κρατών μελών. Και υπάρχει η λογική του reinsuring, όπου υπάρχει μια μεταφορά. Κοιτάξτε σας διακόπτω γιατί θα πρέπει να πάω στη διάσκεψη των Προέδρων, λέει ο κύριος Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ashworth αν ε, θέλει να συνεχίσει την Προεδρία. Ζητώ συγγνώμη. Ε, βρίσκω πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επιλεκτική και εξαιρεί τις μη συνεργαζόμενες σε δικαιοδοσίες νομικές και εννοούμε φυσικά τους φορολογικούς παραδείσους, δηλαδή τις χώρες οι οποίες οργανώνουν την απόκρυψη κερδών κεφαλαίων ε, και ε, που ε, έχουν πάντα την εμπιστευτικότητα των τραπεζικών καθαθέσεων σαν προτεραιότητα. Ευχαριστώ κύριε ο εκπρόσωπος της τράπεζας. Τώρα για τα λεγόμενα asset management. Εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε έναν από τους σκιώδεις. Η Επιτροπή είναι ε, διαθέσιμη να αναλάβει ε, την διαχείριση. Έχουμε τους πόρους να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνει αυτό αν το αποφασίσετε ας πούμε από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου θα εξοικονομηθούν χρήματα. Όχι ότι δεν το κάνει καλά η τράπεζα, αλλά εμείς μπορούμε να το κάνουμε με χαμηλότερο κόστος για την Κούβα. Δεν έχουμε ακόμα εξετάσει την πρόταση της εισηγήτριας για να διευρύνουμε την δράση μας και εκεί. Εδώ επιφυλασσόμεθα. Είμαστε απολύτως ουδέτεροι, θα πρέπει να το ελέγξουμε το θέμα με τους συναδέλφους από της Τράπεζας και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στην Αντιπρόεδρο Μογκερίνη να δούμε ποια είναι η δική τους γνώμη. Θα είναι πολύ πιο ε, ενημερωμένοι από εμά για τέτοιου είδους θέματα. Ή αν θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε την Κούβα σαν πιθανώς επιλέξιμη για το μέλλον. Θα υποστηρίξω επίσης και την θέση των συναδέλφων της τράπεζας σχετικά με, τα, με τις διαδικασίες και τα ε, πρακτικά χαρακτηριστικά των ε, αναγκών δημοσιοποίησης στοιχείων, ίσως τίθενται εδώ το θέμα της εμπιστευτικότητας. Κάποια στοιχεία είναι δύσκολο να ε, δημοσιευθούν. Σαν παράδειγμα εμείς υποστηρίζουμε αυτό το οποίο προτείνετε εσείς για την ισότητα των φίλων, αλλά στις συστηματικές ex post εκθέσεις ε, ε, μη ομογενοποιημένων στοιχείων η άποψή μου είναι ότι θα είναι ε, λίγο δύσκολο να λάβουμε υπόψη μας την προβληματική του φύλου εκεί γιατί πολλές φορές ε, στα πλαίσια των ε, εγγυήσεων που δίδονται είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς το φύλλο του δικαιούχου. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει ε, να είμαστε λογικοί στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουμε τώρα για την καταλληλότητα, την οποία έθεσε το θέμα της καταλληλότητας που έθεσε ο κύριος Σαρτουρί. Εμείς κάνουμε ε, συστηματικές τακτικές εκθέσεις γύρω από αυτό. Η τελευταία έκθεση έγινε στην αρχή του χρόνου. Ε, πιστεύουμε ότι το 9% είναι κατάλληλο, αλλά μιας και διευρύνουμε την κάλυψη των αρμοδιοτήτων μας για να συμπεριλάβουμε και κάποιους νέους τομείς, όπως η κάλυψη του εμπορικού κινδύνου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα μπορούμε να έχουμε αυτό το περιθώριο, τον, την προφύλαξη από το 9 με 10%. στην έκθεση της ΕΦΕΤ. Είναι αλήθεια ότι τα θέματα που προτείνει η ΕΦΕΤ τα συζητάμε. Ίσως να μην γνωρίζετε την ορολογία μας, αλλά το θέμα είναι ότι μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες και η Επιτροπή εξ πόστο μπορεί να ζητήσει να α, διευρυνθεί η κάλυψη. Αυτό ίσχυσε για το FC1 θα μπορούσε να γίνει και για το FC2 αν θεωρήσει το Κοινοβούλιο ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ως προς το πώς ε, εμείς θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την κάλυψη. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάποιο θεωρητικό πρόβλημα αν θελήσουμε να το κάνουμε. Γιατί αυτό θα επιτρέψει εξορισμού ε, την, Ευρωπαϊκή Τράπεζα να επιταχύνει τις διαδικασίες ε, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη αναγκών προσφύγων ε, είναι καλό να λειτουργεί κανείς γρήγορα. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο συναδελφο τον λόγο λοιπόν πλέον για το θέμα αυτό, γι' αυτό θα επιστρέψω στην εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αλλά και την Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά τους. Θα ήθελα να προσπαθήσω όμως να δώσω κάποιες εξηγήσεις λεπτομερέστερες, κάποιες από τις προτάσεις αυτές. Σχετικά με την κατανομή αυτής της αύξησης των πιστώσεων ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες, στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, όπως είπα στην αρχική μου παρέμβαση, και λαμβάνοντας υπόψη την, επιπλέον την έκτακτη προσπάθεια η οποία έχει γίνει για τη Μολδαβία και κυρίως για την Ουκρανία, είναι σαφές ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επενδυτικό και ταυτόχρονα θα ήταν ενδιαφέρον να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις χώρες ε, του Νότου στις οποίες υπάρχουν ε, πάρα πολλοί ε, πρόσφυγες και, τους και οι οποίες υποδέχονται πάρα πολλούς πρόσφυγες. Το να συνεχιστεί ο συσχετισμός αυτός, ο λόγος αυτός ένα προς τρία και να προσπαθούμε με κάποιες μικρές ε, ρυθμίσεις να διατηρήσουμε αυτό το ένα προς τρία θα μπορούσε να είναι σωστό, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές γειτονίας. Ε, δεν είναι εύκολο βέβαια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε παρόλα αυτά περισσότερο τη Λατινική Αμερική. Πρώτον, γιατί έτσι και αλλιώς προτείνεται ε, να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες περιοχές η Κούβα και από την άλλη γιατί νομίζω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Λατινική Αμερική θα πρέπει να ενισχυθεί ιδιαίτερα μετά από τις θέσεις τις οποίες εκφράζει ο Τραμπ ε, για τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ε, γεωστρατηγική την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσπαθήσει να είναι περισσότερο παρούσα γιατί τελευταία έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι το λάθος του Τραμπ να συγκεντρώσει την προσοχή του στην εσωστρεφή αντιμετώπιση ε, της ε, περιοχής αυτής γενικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι μια ευκαιρία για μας. Τώρα ειδικά για την Κούβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Μογκερίνη το Δεκέμβριο του 2016 εξέφρασε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιθυμία να αλλάξει τις σχέσεις τις οποίες έχει α, με την Κούβα. Δεν, αυτό αποφασίστηκε λοιπόν το 2016 δεν έγινε αυτό γιατί το Κοινοβούλιο θέλει να επιβεβαιώσει τη συμφωνία αυτή νομίζω ότι είναι ένα βασικό βήμα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις με την Κούβα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί σαν κατά προτεραιότητα χώρα επιλέξιμη. Είναι επίκαιρο το να συζητιέται τώρα το συγκεκριμένο θέμα, είναι ένα πολιτικό μήνυμα θα έλεγα προς την σωστή κατεύθυνση. Και τώρα για τα 35 εκατομμύρια ε, για την αύξηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κατηγορία 4 έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε αν μπορούμε να βρούμε 35 εκατομμύρια και επιπλέον ποσά για τη χρηματοδότηση των πολιτικών που έχουν σχέση με τους πρόσφυγες. Και θα πρέπει ε, να μπορέσει να βρει αυτή, τα, αυτά τα ποσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς όμως τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά γιατί η πολιτική υποδοχής και πρόνοιας και φροντίδας ε, των μεταναστών ήταν απέσια. Αλλά τουλάχιστον να βρούμε ε, μια συμφωνία για τη συγκεκριμένη κατηγορία Νομίζω ότι με λίγη καλή θέληση θα υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα ποσά αυτά για να βελτιώσουμε την ανάπτυξη των χωρών γειτονίας. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Να υπενθυμίσω και το χρονοδιάγραμμα τροπολογίες 2 Μαρτίου 6 η ώρα το απόγευμα. 19 Μαρτίου, έγκριση της γνωμοδότησης της ΣΥΝΤΑ, ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής μας για τις τροπολογίες 20-21 Μαρτίου, στη συνεδρίαση τότε. Στις 21 Μαρτίου επίσης θα εγκρίνουμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ και ε, στις 24 Μαρτίου έχουμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΜΠΕ. Εμείς ε, θα ψηφίσουμε στις 30 Μαρτίου και 3 Απριλίου στην Ολομέλεια και από εκεί και πέρα εντολή για διαπραγματεύσεις, πρώτος τριμερής διάλογος 10 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και πάλι. Με αυτό ολοκληρώνεται η πρωινή συνεδρίαση, πέρα τη συνεδρίαση και να υπενθυμίσω στους αδέλφους ότι θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα το απόγευμα, εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ.